Chers collègues, nous allons commencer la, la réunion et je vous invite à prendre place. παρακαλώ Merci beaucoup. Je vais commencer. Θα ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στην κυρία Θεοχάρους που έχει μια ανακοίνωση να μας κάνει. Δεν τη βλέπω. Well, dear... Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι η τελευταία μου παρουσία εδώ. Πήγα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και λυπούμε που δεν θα είμαι μαζί σας πια. Ήταν πολύ παραγωγική και έξοχη η περίοδος της κοινοβουλευτικής μου ζωής. Εύχομαι να είμαι μαζί σας την επόμενη θητεία, αν καταφέρω να επανεκλεγώ. Θα είμαι στη διάθεσή σας πάντα και θα συνεχίσω να εξετάζω τα θέματα που συζητούμε. Ο κύριος Πιτσιλίδης θα με αντικαταστήσει εδώ. Είναι νέο μέλος του Κοινοβουλίου από την Κύπρο, αντικαθιστά τον κύριο Κασουλίδη και ελπίζω να είναι καλύτερος από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Κάσμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν ρώτησα την ομάδα μου, αλλά θέλω να πω στην Ελένη, επιφανή, την επιφανή δόκτωρα Θεοχάρους, ότι θα μας λείψετε. Η συνεργασία με όλε τις πολιτικές ομάδες υπήρξε απίστευτη. Υπερασπιστήκατε αρχές, υπερασπιστήκατε τα δικαιώματα των γυναικών και τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολύ συχνά μισητών μειονοτήτων όπως είναι οι λεσβίες, οι ομοφιλόφιλοι, οι φιλομεταβατικοί, ε, θα παραμείνω στη μνήμη μου, ήσασταν υπέροχοι, ισχυροί σύντροφο, σα θυμόμαι πάντα, θυμάμαι πάντα όχι μόνο σαν πολιτική, αλλά σαν προασπίτρια των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σα ευχόμαστε κουράγιο στα νέα σας ε, καθήκοντα και ο κύριος Γκέμιτσεκ θέλει να πάρει το λόγο. Ο Γκέι Μίτσελ. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ την Ελένη για το χρόνο. Ήταν αξιόπιστη. μα βοηθούσε. Εργαζόταν σκληρά η συνάδελφο. Τώρα πηγαίνει σε μεγαλύτερα θέματα, ηγείται τη αντιπροσωπεία τη, θα ηγηθεί τη αντιπροσωπεία τη. Δεν θα τη βλέπουν τόσο πολύ, αλλά ξέρουμε ότι είναι εκεί και θα μα υποστηρίζει. Και πραγματικά θα την ευχαριστήσουμε, θα την ευχαριστήσουμε για τη δουλειά που έκανε, θα μου λείψει σε επικεφαλίστα τη αντιπροσωπεία. Ο κ. Πεσαλίδη που έρχεται δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει, αλλά τα καθήκοντα του Κυπρίου είναι να μας καλεί όλους στην Κύπρο για τις πρώτες δύο εβδομάδες του Αυγούστου. Τη εύχομαι τη Ελένη Τύχη, την ευχαριστώ, θα είναι στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, οπότε θα την βλέπουμε συχνά. Και είναι μεγάλη μας χαρά, ήταν μεγάλη μας χαρά, ε, ήταν ένα από τα όκνα μέλη μας. Ο κύριος Γκέρανς έχει το λόγο. Θα ήθελα πάνω από όλα να ευχαριστήσω τη συνάδελφό μας, που μας υποστήριξε πολύ σε σημαντικές εκθέσεις. Να τις πω απλώ έφυγε. Ε, αλλά θα είναι πάντα εκεί, μπορεί να έρχεται. Ξέρει πάντα ότι υπάρχουν πολλές καινές θέσεις εδώ και μπορούμε να την υποδεχόμαστε. Euh, και εγώ θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμή στην Ελένη, διότι συχνά πήγαμε σε αποστολέ ανθρωπιστικές, μπορούμε να το πούμε έτσι. Η ε, μία μας έκανε να έρθουμε κοντά, διότι η ε, Ελένη παραλίγο να χάσει τη ζωή Παρ' όλα αυτά, πάντα συνέχισε και για μένα είναι μια μεγάλη κυρία και με μεγάλο, μεγάλη συγκίνηση τη βλέπω να φεύγει. Ευχαριστώ. Κατρίν Γκρές. Bien, alors... Η Κατρίν Γκρές. Να προσθέσω και εγώ ε, τους επένους μου, να χαιρετήσω την αναχώρησή σας, την αναχώρησή σου και να πω εν πάση περιπτώσει ότι ανακάλυψα τι άτομο ήσουν πάντα στην τελευταία μας ήρθα στο Στασβούργο, εκείνες τις δύσκολες στιγμές που ζήσαμε όλοι μαζί, τις δραματικές στιγμές που σε είδα να τρέχεις βιαστική ε, για να βοηθήσεις τον ε, αντιπρόεδρο που κατέρευσε ε, και ειδού δεν ήξερα καν ότι ήσουν γιατρό τώρα το ξέρω. Γνωριστήκαμε καλύτερα, καλό θάρρο και πολύ σύντομα, καλό κουράγιο. Σύντομα στο πολιτικό μέλλον θα συναντηθούμε. Ο κύριος Ντέβα επίσης. Και εγώ θα ήθελα να πω πόσο θα μου λείψει η Ελένη, ρητωμένη, ε, καλή, ε, γενναιόδορη, ε, ε, ε, είχε μεγάλη ευφράδια, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάντα περιστατωμένα οι γνώσει τη και ξέρω θα τα λέμε αλλού. Με όλα αυτά λοιπόν, Ελένη φεύγεται με άριστο τρόπο για τα νέα καθήκοντα. Θα προβούμε στη ψηφοφορία. Η πρώτη ψηφοφορία μας. On doit Πρέπει να κάνουμε μια δοκιμή να δούμε αν λειτουργούν οι κάρτε μου, λέει η γραμματεία. Έχετε όλοι τι κάρτε σα. Ο κ. Κάσμαν δεν έχει τη δική του. Προσπαθούμε λοιπόν, κάνουμε δοκιμέ. <laughs> bon, le vote est ouvert. Ξεκινάει η δοκιμή λοιπόν. Ψηφίζουμε. Μα Μας λείπουν δύο ψήφοι. Α, εγώ δεν ψήφισα. Ναι. Και του κύριου Κάσμαν, οι άλλοι εντάξει, καλά είμαστε. Ο κύριος Κάσμαν δεν έχει. Δουλεύει. 24 κάρτες λοιπόν, βλέπω. Πέρας ψηφοφορίας. Ωραία, τέλεια. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροποποίηση της Συμφωνίας Κοτονού της 23ης Ιουνίου 2002, έκθεση Κάσμαν, δεν υπάρχει τροπολογία, ψηφίζουμε λοιπόν την έκθεση ως έχει, ψηφίζουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται Α, ναι, τώρα έχουμε πέρας ψηφοφορίας. 24 ψήφοι υπέρ, ομόφωνα. Εγκρίνατε. Και τώρα θα ψηφίσουμε συμφωνία σύμπραξης οικονομικής με την Κεντρική Αφρική. Έκθεση της Τζουτίθ Αργεντίνη. Ψηφίζουμε τώρα τις ε, τροπολογίες. Ψηφίζουμε την ομαδικά την τροπολογία 2, 3 και 4. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Εν συνεχεία η τροπολογία 1 έχει αποσυρθεί. Τελική ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος, ηλεκτρονική επαλήθευση θα γίνει. Ξεκινάει τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκαεπτά ψήφοι υπέρ. Τρεις ψήφοι κατά και τέσσερις αποχές. Και αυτό αποτελεί το τέλος ε, των ψηφοφοριών. Πάμε τώρα στο σημείο 15, 15 της ημερήσιας ε, διάταξης. Η στόχοι της χιλιετίας, οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας. Θα καθορίσουμε το πλαίσιο που θα ακολουθήσει το 2015. Έχουμε ξεκινήσει την επεξεργασία του θέματος. Ο κύριος Κασμάρεκ έχει συντάξει μια έκθεση και θα ήθελα να προβώ σε κάποιες γενικές παρατηρήσεις πριν του δώσω το λόγο πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή ο οποίος δεν έχει έρθει ακόμα. Α, εσείς, μάλιστα. Όπως γνωρίζετε, το Σεπτέμβριο φέτος θα διεξαχθεί στο ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη μια ειδική εκδήλωση που θα αποτιμήσει τις προσπάθειες που έχουν γίνει για να επιτευχθούν οι στόχοι της χιλιετίας. Συζητήθηκαν οι προσπάθεια που να γίνουν να μέχρι το 2015, η μορφή και οι στόχοι του μελλοντικού πλαισίου. Οι δεσμεύσει που ελήφθησαν στη σύσκεψη του Ρίο ΣΥΝ του Ιουνίου του 2012 θα πρέπει να εφαρμοστούν. Άρα θα χρειαστεί να παγιωθεί η δουλειά που έχει γίνει σε αυτή τη διάσκεψη Ρίο ΣΥΝ και μέσω της ομάδας εργασίας της ανοιχτής ε, έγιναν οι προσπάθειες συζητήσεις, θα πρέπει να προσπαθήσει να συμμετάσχει η διεθνή προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση και να συμβάλλει συντονισμένα και συγκεκριμένα στην προσπάθεια. Όχι μόνο στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και εντός άλλων διεθνών βημάτων. Θα πρέπει να ξεκινήσει επικοδομητικό διάλογο η Ευρωπαϊκή Ένωση με όλου τους συμμετέχοντες, να προσπαθήσει να πετύχει ευρεία συνένεση και να υπάρξουν σαφείς συνεισφορές και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για να είναι φιλόδοξο το αναπτυξιακό πρόγραμμα. Θα πρέπει αμέσως όμως να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το γενικό πλαίσιο της εκθέσεώς του. Ο κύριος Γκί Μίτσελ, αντιαπουσία του κυρίου Γκασμάρεκ, θα παρουσιάσει την έκθεσή του. Ο κύριος Γκάι Μίτσελ, λοιπόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δυστυχώ ο Φίλιπ δεν μπορεί να είναι μαζί μα σήμερα, γιατί είναι πολύ βαριά κρυωμένο και δεν μπόρεσε να ταξιδέψει. Ε, θα προσπαθήσω εγώ να σα δώσω μια γενική εικόνα των σημείων και των προτάσεων που περιλαμβάνονται στην έκθεση, στο σχέδιο έκθεση μάλλον του Φίλιπ. Την τελευταία δεκαετία οι στόχοι της χιλιετίας έχουν ε, βοηθήσει στην εξέλιξη της ε, φτώχειας και την περαιτέρω ανθρώπινη ανάπτυξη. Έχει υπάρξει κάποια πρόοδος και είναι σημαντικό να την αναγνωρίσουμε, όχι για κανένα λόγο, αλλά για το ότι ανησυχούν ε, οι πολίτες μας και δεν θα, συνεχίσουν να μας στηρίζουν εάν δεν ξέρουν ότι έχει γίνει κάποιο είδους πρόοδος. Βεβαίως υπάρχουν πάντα προκλήσεις που πρέπει να λυθούν και φυσικά υπάρχουν πράγματα που ακόμη πρέπει να γίνουν. Όπως είπατε Πρόεδρε, το, σεπτε... το φθινόπωρο του τρέχοντος, του ε, προηγούμενου του μάλλον, Συγγνώμη, τον Σεπτέμβρη του 2013 θα ε, υπάρξει μια διάσκεψη η οποία θα προσπαθήσει να κάνει μια εκτίμηση της κατάστασης ε, και, πώς, ε, και θα μελετήσει το πώς μπορούν να επιτευχθούν οι ε, στόχοι μετά το 2015. Υπάρχει και το Ρίο όπου η διεθνής κοινότητα συμφώνησε να, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις για τη βιωσιμότητα και ξεκίνησε την διαδικασία για την δημιουργία των στόχων για, τους βιώσ, για τη βιώσιμη ανάπτυξη που θα προωθηθούν από τον ΟΗΕ και την ανοιχτή ομάδα εργασίας τους. Να σας θυμίσω επίσης ότι ε, στις 27 Φεβρουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε κάτι πολύ σημαντικό με τίτλο «Μια αξιοπρεπή ζωή για όλους. Τέλος στη φτώχεια και, και ένα βιώσιμο μέλλον για τους πολίτες». Ε, κάποιοι είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον Επίτροπο Πίμπαλξ αρκετά έντονα και θα συμφωνεί η Επιτροπή σας το έγγραφο αυτό τη Κομισιόν περιλαμβάνει πολύ σημαντικέ προτάσεις και κατευθυντήριε γραμμέ, ώστε να υπάρξει ένα ένας τρόπο τρόπος και μια ολοκληρωμένη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση μετά το 2015. Παρ' όλα αυτά, βεβαίω θα πρέπει να περιμένουμε κάποιες προσαρμογέ για την κατάσταση αυτή την Άνοιξη θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε μια κοινή θέση για την Ευρώπη για τέτοιε διεθνεί ε, διαδικασίε και δραστηριότητε. Η κοινή προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι απαραίτητη μέχρι τα μέσα του τρέχοντο έτου. Η έκθεση λοιπόν είναι η πρώτη. Ε, ε, το πρώτο βήμα σε επίπεδο Κοινοβουλίου μετά το Ρίο και σε διεθνές επίπεδο και με την, ε, με την προοπτική να αναθεωρηθούν οι στόχοι της χιλιετίας ε, για το μετά το 2015. Ε, η εξάλληψη της φτώχειας και η επίτευξη των, της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να είναι η τομής προτεραιότητα στο νέο πλαίσιο, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό που ονομάζουμε αξιοπρεπή ζωή για όλους. Όπως αναφέρεται στο αποτέλεσμα της διάσκεψης Ριωσινή 20, το, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δει την υγεία και την εκπαίδευση ως, βασικά, ως βασικούς τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης και ως κινητήριες δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης. Για να μπορέσουμε λοιπόν να εξαλείψουμε τη φτώχεια και να εξασφαλίσουμε την επιστηστική ασφάλεια, πρέπει πρώτα να επιτύχουμε το στόχο της, ε, του καθορισμού ε, προτύπων για, την, για το καθαρό νερό, για την ε, διατροφή, και επίσης θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στην αντιμετώπιση ε, μη μεταδιδόμενων νοσημάτων όπως ο καρκίνος. Έτσι προτείνει ο εισηγητής. Η διάσκεψη 2 συν 20 ξεκαθάρισε ότι για να επιτύχουμε τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη χρειαζόμαστε θεσμικά όργανα σε όλα τα επίπεδα τα οποία θα είναι διαφανή, θα είναι δημοκρατικά, επομένως χρειάζεται σαφής δέσμευση ε, για δημοκρατική διακυβέρνηση και αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο νέο πλαίσιο. Για να επιτύχουμε το στόχο αυτό πρέπει το Κοινοβούλιο να παίξει ένα σημαντικό ρόλο έτσι ώστε να θεωρήσει κτήμα του αυτέ τι ε, πολιτικέ ε, βιώσιμη ανάπτυξη, να κάνει ε, συζητήσει για το θέμα αυτό και να δεσμευθεί για δράσεις για του τομεί αυτού και βεβαίω όλα αυτά να περάσουν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκής αλλά και Διεθνού νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε την όλη διαδικασία έτσι ώστε και οι αρχέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και οι στόχοι της για την βιώσιμη ανάπτυξη να μπορούν να επιτευχθούν. Στην έκθεση επίσης αναφέρεται και η ειρήνη, η ασφάλεια και η ανάπτυξη. Οι ένοπλες συγκρούσεις και οι καταστάσεις μετά την, ε, τις σειράξεις εξακολουθούν να αποτελούν ε, ε, πρόσκομα για την ε, ανάπτυξη. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι ζουν σε περιοχές που βρίσκονται σε, εμπόλεμες κατάστα... σε, εμπόλεμες... Ε, σε εμπόλεμη κατάσταση και δεν... αυτό βεβαίως δεν μπορεί να σημαίνει επιτυχία των στόχων της χιλιετίας. Συνάδελφοι, οι στόχοι της, ε, για τη βιώσιμη ανάπτυξη ε, περιλαμβάνονται στην έκθεση μέσω συγκεκριμένων προτάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει την χρήση συγκεκριμένων ε, στόχων για την ενέργεια, για το νερό, για τη βιώσιμη χρήση της γης, για την ε, επάρκεια των πόρων, την προστασία των θαλάσσιων πόρων, αλλά και τη βιοπικιλότητα. Για την κατανομή των κονδυλίων, η έκθεση τονίζει τη σημασία της, ε, μιας συζήτησης ε, για την πολιτική ε, που θα συμπεριλαμβάνει όλους τους τομείς και τους στόχους για την βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015. Ο κύριο Κάτσμαρκ επίση τονίζει την ανάγκη για βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων μηχανισμών βοήθεια αλλά και των δωρητών για την ανάπτυξη τροποποίηση των φορολογικών πολιτικών ε, με αποτελεσματικούς φορολογικούς μηχανισμούς, ενίσχυση των ιστορικών εσόδων μέσω αποτελεσματικής φορολόγησης και αντιμετώπιση της διαφθοράς, καθώς επίσης και ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Τώρα, για τους υποπτικούς μηχανισμούς και τους δείκτες, η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία σαφών και ξεκάθαρων δικτών, έτσι ώστε να μετράτε η πρόοδος, να προωθείτε η λογοδοσία, να αυξάνετε η ευαισθητοποίηση και να, τονίζετε, ε, να τονίζονται οι πρακτικές αναχώρα. Επίσης, η έκθεση θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι υπηρεσίες του ΟΗΕ αλλά και οι διεθνείς οργανισμοί θα πρέπει να προχωρήσουν σε ένα κατάλληλο μείγμα ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων για την μέτρηση και των δικτών. Ε, επίσης, ένας πολυδιάστατος μηχανισμός θα πρέπει να μπορεί να αξιολογήσει και να μελετήσει τα σχετικά θέματα, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η φτώχεια, η ανισότητα, η ισότητα των φύλων και η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής βοήθειας. Η συνεκτικότητα των πολιτικών για την ανάπτυξη και ο συντονισμός μεταξύ των δωρητών είναι ένα ζωτικό στοιχείο για ε, να υπάρξει μια συντονισμένη ευρωπαϊκή θέση. Είναι λοιπόν ζωτική σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει υπόψη της τους στόχους ε, για την ε, αναπτυξιακή συνεργασία σε όλους τις πολιτικές και να εφαρμόσει σε όλε τι πολιτικές μάλλον που εφαρμόζει και που μπορεί να ε, επηρεάσουν τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Κλείνοντα κυρία Πρόεδρε, να αναφέρω κάποιες αρχές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον ορισμό το της και συνεκτικής ευρωπαϊκής θέσης, έχοντας ως στόχο τις διαπραγματεύσεις για το νέο αυτό πλαίσιο. Θα πρέπει να βασιστούμε στις επιτυχίες που έχουμε ε, καταφέρει μέχρι τώρα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε βεβαίως τις νέες παγκόσμιες προκλήσεις. Η μελλοντική ατζέντα θα πρέπει να είναι ε, φιλόδοξη, συνολική, πολυδιάστατη και ευέλικτη θα πρέπει να έχει ε, στόχο να λύσει προβλήματα σε χώρες που θα, με συγκεκριμένους ε, τρόπους ανάλογα με τις ανάγκες τους και βεβαίως θα έχει μετρήσιμους στόχους. Η κατάσταση μετά το 2015 θα πρέπει να βασιστεί σε αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητας, μη διακριτικής μεταχείρισης, βιωσιμότητας, καλής διακυβέρνησης και ε, συνεκτικότητας των πολιτικών για την ανάπτυξη με το στόχο να δημιουργηθεί ένας δίκαιος και βιώσιμος κόσμος όπου ο καθένας μπορεί να εξασκεί τα δικαιώματά του και να ζει ελεύθερος από τη φτώχεια. Πρέπει να κινητοποιήσουμε όλους τους πιθανούς οικονομικούς πόρους και, καθώς και όλα τα καινοτόμα, όλους τους καινοτόμους οικονομικούς μηχανισμούς για το νέο αυτό πλαίσιο. Εκ μέρους του εισηγητού, λοιπόν, ε, προτείνω αυτή την ε, έκθεση στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. <coughs> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γκέι Μίτσελ που μας παρουσίασε την έκθεση του κύριου Κάτσμαρεκ. Είναι ένα σαφές περιεκτικό σχέδιο έκθεσης, ευανάγνωστο, σαφές και περιεκτικό. Θέλω να ευχαριστήσω και την ε, Επιτροπή για μια φιλόδοξη ε, και ευρή ανακοίνωση στην οποία αναφέρθηκε ο Γκέι Μίτσελ. Είχα το προνόμιο και εγώ να συζητήσω το θέμα αυτό με τον Επίτροπο Πίμπαλξ, με εσά μαζί κυρία Πρόεδρε και άλλου συναδέλφου. Αυτό το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι ότι το Συμβούλιο έχει να κάνει τώρα τη δουλειά. Δηλαδή ουσιαστικά να συμφωνήσουν 27 μεταξύ τους και έπειτα να συμφωνήσει το Συμβούλιο με Κοινοβούλιο και Κομισιόν ώστε να μιλήσουμε με μια φωνή για το θέμα αυτό διότι αν Είμαστε κατακαιρματισμένοι. Ουσιαστικά ε, υπονομεύουμε αυτό τον ακρογωνιαίο λίθο και κυρίως ε, αυτοί που θα πληγούν είναι οι ε, φτωχότεροι. Το Σεπτέμβριο λοιπόν θα πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή για να καταφέρουμε να πετύχουμε αυτούς τους πολύ φιλόδοξους στόχους. Ο κύριος Μίτσελ αναφέρθηκε στην έκθεση του κύριου Κατσμάρε και στο θέμα και στη σημασία που έχει το ζήτημα. Αμερική, Ασία, Λατινική Αμερική. Πολλές ιστορίες που ακούμε σήμερα από αυτές τις υπήρους είναι ιστορίες επιτυχίας και προόδου. η στόχοι της χιλιετίας, οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας είναι επιτυχία. Και πρέπει να το τονίσουμε αυτό αν θέλουμε τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν έτσι περαιτέρω. Στο φιλόδοξο μονοπάτι που έχουμε να διανύσουμε προς τα εμπρός. Όπως γνωρίζετε πολλά άλλαξαν μετά την έγκριση του σχεδίου για τους αναπτυξιακούς ε, στόχους. Μετά είχαμε τη συμφωνία Glen Eagles. Πολλά άλλαξαν. Είχαμε οικονομική ύφεση. Πολλές χώρες ε, είναι απρόθυμες ε, το 0,7 του ΑΕΠ να το συνεισφέρουν, κάτι απαραίτητο. Τώρα όμως πρέπει να διδαχθούμε από τα μαθήματα του παρελθόντος. Πρέπει να αναλύσουμε τι δεν καταφέραμε να κάνουμε σωστά ή μάλλον να καταλάβουμε τι κάναμε καλά και να είμαστε ειλικρινεί για το τι δεν κάναμε καλά. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε του γλίσχρου πρόσωπου που έχουμε στη διάθεσή μα να του ε, διαθέσουμε ε, σε αποτελεσματικέ ε, στρατηγικέ για τη μείωση τη φτώχεια. Το πλαίσιο γενικώ των αναπτυξιακών στόχων και οι στόχοι περιβιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να ειδωθούν ως ένα κοινό, μια κοινή δέσμη στόχων. Ανθρώπινη ανάπτυξη επίσης, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο, σε ένα μάλλον περιβάλλον, ε, πάρα πολύ ε, σημαντικά και αυτά και διασυνδεδεμένα μεταξύ τους στοιχεία. Είναι σημαντικά για μας ως βουλευτές. Σε ό,τι αφορά την καθολική εφαρμογή του μελλοντικού πλαισίου και εγώ θέλω να υπάρχει συνολική ευθύνη, είναι σημαντικό επίσης η ε, στόχη να είναι περιορισμένη στον αριθμό. Ίσως όμως ε, θα μπορούσαμε να έχουμε διαφορετική στρατηγική για κάθε χώρα. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, κάτι που θα, προσπαθήσουμε, να το ταιριάξουμε σε όλους, ε, one size fits all, κάτι που είχαμε εφαρμόσει με αποτυχία στο παρελθόν. το θέμα είναι ότι και η υγεία, η αναπτυξική στόχη της χιλιετίας για την υγεία πρέπει να παρέμει προτεραιότητα. Δεν έχουμε επιτύχει επαρκή πρόοδο. Επίσης αυτό περιλαμβάνει τα σεξουαλικά αναπαραγωγικά δικαιώματα. Είναι συνιστόσα της υγείας αν θέλετε, είναι ο δρόμος για την υγεία. Θα πρέπει λοιπόν να τα πούμε πιο ε, ξεκάθαρα και να, να είμαστε και ενιαίοι, γιατί ε, αν παραμείνουμε σιωπηλοί θα είναι καταστροφή ε, για πολλούς άνδρες και πολλές γυναίκες. Το κάναμε αυτό πέρυσι και για το, στο πλαίσιο του ΕΕ θα είναι καταστροφικό αν το επαναλάβουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ξέρω ότι δέχεται επιθέσεις για τον ηγετικό ρόλο που τήρησε αυτή την περίπτωση. Μιλώντας για τη δική μου ομάδα, αλλά και άλλοι πιστεύω, ε, στηρίζουμε εμείς ε, ε, αυτή την προσπάθεια και τη στηρίζουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Επίσης, τη διάσταση της ισότητας πρέπει να τη συμπεριλάβουμε στους ανάπτυξες της χιλιετίας. Και τέλος, την ε, ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή πρέπει να είναι η βάση, το θεμέλιο για την ε, δουλειά μας. Έχω επίσης και κάποια άλλα σχόλια, αλλά νομίζω ότι θα τα αφήσω για τη συζήτηση σε μεταγενέστερο στάδιο. Είναι φιλόδοξο το σχέδιο, είναι εκτεταμένο, ε, αλλά θα πετύχει μόνο αν έχουμε και τη δέσμευση των πόρων. Αν δεν έχουμε το 0,7 του εθνικού καθάριστου εισοδήματος, Είπαμε ότι αυτό είναι απαραίτητο και αν δεν έχουμε και την πρόσθετη αυτή χρηματοδότηση που συζητήσαμε, ουσιαστικά θα έχουμε μόνο ε, μια τρύπα στο νερό και αυτό δεν θα βοηθήσει σε τίποτα. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντόνσκης. Um, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την συμβολή μας ε, για αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να σας πω ότι η γνώση, η εμπειρία, η τεχνογνωσία είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να το μοιραστούμε με τις αναπτυσσόμενες χώρες και από αυτό το πρίσμα νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε και την εμπειρία που θα μπορούσαμε να μεταλαμπαδεύσουμε. Τα κράτη της Κεντρικής, Ανατολικής Ευρώπης, οι χώρες της Βαλτικής έχουν τέτοια εμπειρία. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν και πολλές χώρες που είναι σε διαδικασία μετάβασης προς τη δημοκρατία, προς την ε, οικονομία της ελευθερής αγοράς, ε, τα ίδια τα βλέπουμε και σε άλλες χώρες αναδυόμενες και γι' αυτό χρειάζεται να υπάρξει ε, η εμπειρία αυτή από τις χώρες μετάβασης και την έχουν αυτή την εμπειρία πολλές χώρες. Οι χώρες της Βαλτικής, κεντρικές, Ανατολ... χώρες κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ήταν μια ιστορία επιτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι σημαντικό. Μπορεί να αντλήσουν διδάγματα από αυτή την επιτυχία οι αναπτυσσόμενες χώρες. Και δεν νομίζω ότι μόνο τα οικονομικά ισχυρά κράτη-μέλη τη Ένωση θα πρέπει να συνεισφέρουν στην ε, αναπτυξιακή πολιτική, αλλά όλα τα μέλη, ακόμη και η Βαλτική, τα κράτη τη Βαλτική. Δεν είναι μόνο μια πολιτική και ηθική υποχρέωση, είναι καθήκον όλων των κρατών μελών. Και τέλο, ήθελα να τονίσω ότι εν καιρό χρηματοοικονομική κρίση οι πόροι, ηλικοί και μη, είναι όλοι απαραίτητοι. Γι' αυτό και αυτή η εμπειρία που επαναλαμβάνω από ε, περίοδο μετάβαση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύτιμη. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Τέιλορ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Κατσιμάρη και ελπίζω να ξεπεράσει το κρεολόγημά του πάρα πολύ σύντομα. Η έκθεσή του νομίζω είναι καλοδεχούμενη. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα με τα οποία κανείς θα μπορούσε να διαφωνήσει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να τονίσουμε ότι η αναπτυξιακή στόχη της χιλιετίας να μην ήταν επιτυχία, γιατί έβαλαν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στην ανάπτυξη, ε, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ε, αρκετά... Ε, το, η εστίαση στη βοήθεια είναι λίγο περιοριστική. Και ιδίω όταν μειώνεται η χρηματοδότηση και τα εφάσματα και οι ροές από ιδιωτικά ιδρύματα και μέσα των άμεσων ξέρων επενδύσεων έχουν διευρυνθεί, έχουν αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο. Νομίζω ότι είναι γι' αυτό άκρο σημαντικό να εστιάσουμε περισσότερο ε, σε μια συνεκτική πολιτική για την ανάπτυξη. Πρέπει να αφήσουμε προοπτική, ε, να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, όπου το διεθνές εμπόριο, το περιβάλλον και η διεθνής χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική να θεωρούνται να εννοούνται ως μια παγκόσμια πολιτική ε, και η διακυβέρνηση βέβαια είναι ένα συστατικό αυτού του θεματολογίου του αναπτυξιακού. Με εστίαση, παραλαμβάνω, στην συνεκτικότητα της πολιτικής για την ανάπτυξη. Θα πρέπει να επεκτείνουμε ε, την, ε, το θεματολογιό μας για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και να καλύψουμε δράσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη. Αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης. Βλέπετε, άκουσα ότι μιλάω, και μπήκαν όλοι μέσα. Υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο είναι κάτι που πονομεύει τις επιτυχίες και τα επιτεύγματα αυτών των απτυξιακών στόχων της Λιτίας πόροι που είναι περιορισμένοι, ε, η ανισότητα, όλα αυτά θα δινωθούν, θα οξυνθούν αυτά τα προβλήματα και ενδέχεται να οδηγήσουν και σε καταστάσεις σύγκρουσης, ανασφάλειας, αβεβαιότητας, βίας, πείνας. Όπως είπε και ο κύριος Κάσμαν, πρέπει να δώσουμε έμφαση στην υγεία. Υπάρχουν ε, νόσοι προβλέψιμες ε, μεταδοτικές που είναι οι άσημες και πρέπει να τις θεραπεύσουμε. Πρέπει να βρούμε την πολιτική βούληση και να έχουμε και την αναπτυξιακή ατζέντα που θα με την οποία θα επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Ξέρετε, πάντοτε με εκπλήσει όταν ακούω να γίνεται λόγος ε, για την ε, ποιότητα ε, της ίδρευσης και της αποχέτευσης, της, την ανάγκη για καλό πόσιμο νερό. Εδώ δεν αναφέρεται και είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό του αναπτυξικού προπολογισμού τη Ένωση που απευθύνεται σε αυτό το στόχο. Άρα, νομίζω ότι αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει νέου στόχου, ώστε να έχουμε έναν εξορθολογισμό τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και βέβαια θα πρέπει να ξεπεράσουμε μια απλή μέτρηση ε, ποσοτικών ή ή ποιοτικών στόχων με βάση το, ε, το θα πρέπει να δούμε το οικολογικό αποτύπωμα. Για παράδειγμα, άλλοι δείκτε πρέπει να χρησιμοποιηθούν επίση. Και αυτοί οι στόχοι, όπω είναι αυτή τη στιγμή, δεν αντιμετωπίζουν ε, τι βασικέ αιτίε τη φτώχεια. Γιατί οι πιο πολλοί φτωχοί, ξέρετε, που ζουν σε χώρε με μεσαίο εισόδημα, όλα αυτά ε, θέτουν ερωτήματα, ε, γύρουν ζητήματα για το μοντέλο τη οικονομία των χωρών αυτών που φαίνεται να αποτυγχάνει, να μην μπορεί να φέρει αποτελέσματα, να μην μπορεί να φέρει ισότιμη ανάπτυξη, ευημερία και υγεία για τους κατοίκους αυτών των χωρών. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω σε σχέση με τα τρόφιμα την ακρόαση που είχαμε τον Ιανουάριο στην Επιτροπή μας. Ακούσαμε αυτή τη μηδενική πρόκληση, ε, ε, πρόκληση μάλλον για τη μηδενική φτώχεια. Είναι μεγάλη πρόκληση. Ο Μπαν Κιμούν ο ΓΓ του ΟΗΕ μιλάει και για μηδενικά απόβλητα τροφών, κατάλοιπα. Θέλουμε να εγγυηθούμε ε, το, τα τρόφιμα, την πρόσβαση ε, των ανθρώπων που τα χρειάζονται στα τρόφιμα. Πρέπει να κάνουμε επενδύσεις στη Γεωργία. Όλα αυτά τα μηνύματα πρέπει να περάσουν και στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο. Πρέπει να ηγηθούμε εμεί τη όλη συζήτηση. Και έχω σχεδόν ολοκληρώσει στην ακρόαση του Ιανουαρίου επίσης που κάναμε. Ακούσαμε και λόγια δυσαρέσκεια από κάποιου εκπροσώπους των τσόμενων χωρών, των δικαιούχων δηλαδή, των αποδεκτών της ε, ανθρωπιστική βοήθειας που λένε ότι δεν είναι ε, αυτό που ε, πιστεύουν οι αναπτυσσόμενες, ή αναπτυγμένες χώρες, αυτό που εμείς οι αναπτυσσόμενες χρειαζόμαστε, αυτό που για μας είναι καλό. Και ήταν ε, πολύ θετικό το μήνυμα. Και θα πρέπει να τα λάβει υπόψη και ο ΙΑ από βλέπω τα λαμβάνει υπόψη όλα αυτά. Τέλος ακούσαμε τον Ιανουάριο Um, and you know particularly in reference to the the the, uh, the για την ανάπτυξη δόση χιλιτίας διάφορα ε, σε σχέση με τους δείκτες και τα λοιπά και ότι υπολογίζουμε με βάση το ΑΕΠ. Μπορεί να μην πετύχαμε τα πάντα. Το θέμα είναι ότι ουσιαστικά η κοινότητα των πολιτών πίεσε τις κυβερνήσεις είπε ορίστε αυτά θέλουν ε, τα Ηνωμένα Έθνη να πετύχουμε, κάντε ό,τι μπορείτε. Άρα έχουν, έχουν χρήσιμότητα, έχουν αξία. Δεν, δεν είναι κακό να προσπαθεί κανείς να πετύχει το καλύτερο και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω μια μορφή ε, μια ομάδα σπουδαστών που ήρθαν εδώ και να θα παραστούν στη συνεδρίασή μας, τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ ελέγχουμε το πώς χρησιμοποιούνται περίπου 54 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και συζητούμε τα κριτήρια τα... και τους στόχους για ε, την επίτευξη των οποίων θα χρησιμοποιηθούν αυτές αυτή οι πόροι, τους στόχους χιλιετίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που βλέπω από το γυμνάσιο, είστε, δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ce sont les élèves de Mirande dans le Gers, un des meilleurs endroits pour vivre en France. De Mirande <laughs> Ok. Viennent de lycée agricole. Από το γεωργικό Λύκειο του Μιράντε, έρχονται από τη Γαλλία. Δεν θα φάνε λοιπόν ε, σήμερα πάπια και δεν θα χάψουν όλα όσα λέμε εμείς. Το ελπίζω. Να προσθέσω αυτά που έλεγε ο Γκάι Μίτσελ. Έξοχη είναι η έκθεση. Σημαντικότατη. Θέτει τα θεμέλια για τη συζήτηση για το ποιο πλαίσιο θα χρησιμοποιήσουμε μετά το 2015. Τι θα κάνουμε στι αναπτυσσόμενες χώρες. Ποιο θα έπρεπε να είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο νέο τοπίο των νέων δωρητών, ιδιωτικών δωρητών όπως το Ίδρυμα Bill Gates που έχει περισσότερα χρήματα από ότι πολλά μεμονωμένα κράτη-μέλη, κράτη-μέλη σε αυτό το νέο τοπίο αναδειωμένων οικονομιών που έχουν ρόλο να παίξουν στις αναπτυσσόμενες χώρες και στη σχέση που θα έχουμε τις χώρες. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Πρέπει να επανεξετάσουμε ποιο θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών, κυρίως των παρόδο, των Ηνωμένων Πολιτειών και των φορέων του ΟΗΕ. Πού έγκυται η προστιθέμενη αξία των παραδοσιακών δωρητών σε σχέση με τους νέους δωρητές. Πολύ σημαντικό θέμα. Χρησιμότατη η έκθεση για τη διεξαγωγή της συζήτησης και θέλω να διαβιβάσω μια ανησυχία μου. Ποια είναι η ανησυχία μου. Από τη μία, κατά την άποψή μου, η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τις αναπτυσσόμενες χώρες έγκυται στο ρόλο που μπορεί να παίξει σαν πολιτικός φορέας που θα τονίσει την ανάγκη που υπάρχει για το σεβασμό των καθολικών αξιών, μη διάκρισης, διακυβέρνησης, ίσων ευκαιριών, βιώσιμης ανάπτυξης Καθολικέ αξίε που θα πρέπει να υποστηριχθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. το κάνει η Κίνα για μα για την ώρα. Αργότερα ναι, είμαι αισιόδοξο. Η Ινδία επίση δύσκολο θέμα. Αλλά αυτό είναι ο ρόλο ο συγκεκριμένο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι ο πειρασμό, Να προχωρήσουμε του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όλα καλά και άγια. Και ο πειρασμό είναι να τονίσουμε την ασφάλεια των τροφίμων, κάτι που είναι πολύ σημαντικό αλλά ίσως ακολουθήσουμε τεχνοκρατική αναπτυξιακή προσέγγιση που θα υπογραμμίζει τεχνικές για τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής, τεχνικές για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, μείωση των συνεπιών κλπ. Πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά. Χρειαζόμαστε βιώσιμη ενέργεια και το καλό για το φαγητό και την ενέργεια είναι ότι είναι πράγματα προσμετρήσιμα μετρήσιμες πτυχές της ανάπτυξης λιγότερη μετρήσιμη είναι η δημοκρατία, σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων κλπ. Ποιο είναι ο πειρασμό, ότι το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κινηθούν προ την ενέργεια, τα τρόφιμα για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά θα λησμονήσουν την μοναδική προστιθέμενη αξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών αυτή, δηλαδή να μεριμνήσουν ώστε αυτές, αυτή η ανάπτυξη θα συνοδεύεται από ανάπτυξη και πρόοδο ανθρώπινα δικαιώματα και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ποιο είναι το πρόβλημά μα. Οι τεχνοκράτε, που είναι ευπρόσδεκτοι και σημαντικοί, θα πρέπει αυτό να το κατανοήσουν. Η ασφάλεια των τροφίμων και ο σεβασμό των μικρών γεωργών ποτέ δεν θα επιτευχθεί χωρί το σεβασμό τη δημοκρατία, χωρί τη συμμετοχή των φτωχοτέρων που θα εισακούγονται στι πρωτεύουσε. Χωρί αυτά δεν θα διαφυλαχθούν οι καθολικέ αυτέ αξίε. Και δεν θα πλησιάσουμε καν στο σεβασμό των και την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Θέλω να αποφευθεί ο κίνδυνος αυτός, δηλαδή να μεληθούν αυτές οι πτυχές. Η μοναδική προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα ήθελα η συζήτησή μας να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση και γι' αυτό σαν βάση είναι έξοχη αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκέραντς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, για εκείνους που ήδη έχουν παραστεί σε αυτού του είδους συνόδους ε, κορυφής θα θυμούνται ότι συναντούν ε, σε ανθρώπους που έχουν μοναδική επιδεξιότητα να λένε κοινοτοπίες. Για να αποφύγουμε η διάσκεψη της Νέας Υόρκης επικείμενη να γίνει κάτι τέτοιο παρόμοιο θα πρέπει να ε, σκεφτούμε τη θέση που θα έχει το Κοινοβούλιο στην όλη συζήτηση. Η υλοποίηση των στόχων της χιλιετίας, των αναπτυσιακών στόχων, χρονολογείται από 15 χρόνια. Έχει ξεκινήσει από 15 χρόνια. Πρέπει να κρατήσουμε τα όσα δούλεψαν και να δούμε τι απέτυχε επίσης. Πρέπει να είμαστε σαφέστατοι. Και εκείνοι θα πρέπει να πούν ότι θα πρέπει να ακουστούν φωνές για να κάνουμε ανάλυση της συνείδησης της Ευρώπης. Να δούμε τι έκανε η Ευρώπη και να δούμε ποιες ευθύνες πρέπει να υπομισθούν και οι άλλοι συνυπεύθυνοι για τυχόν αποτυχίες. πρέπει να εξετάσουμε την τελευταία 15 ετία. Ποια είναι η κατάσταση στις πιο χωρημένες χώρες, ποιες για τις άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, ποια η κατάσταση με τις, για τις χώρες με το μέσο εισόδημα, ποιο σημείωσε πρόοδο, ποιο ο ρόλος του εμπορίου στην εξάλληψη της ένδυας, κάτι που ίσως υποτιμούμε, ίσως να το υπερεκτιμούμε, θα πρέπει όμως να γίνει ένας απολογισμός των ε, μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και πώς ε, επηρέασαν την παρούσα κατάσταση πριν τοποθετηθούμε επί των υπολείπων. Αυτός που πρέπει να παίξει βασικό ρόλο σε όλα αυτά είναι ο Πίμπαλξ. Ήταν αποφασισμένος, τον είδα αποφασισμένο περισσότερο από ποτέ. Πρέπει να τον υποστηρίξουμε. Και Ήμουν ανάμεσα αυτούς που ε, συμμετέχει στην προετοιμασία της συνεδριάσεως. Εμείς θα πρέπει να το υπενθυμίσουμε, να υπενθυμίσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους άλλους εταίρους, κυρίως τους βουλευτές, που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτά που προανέφερα. να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι των αποτυχιών. Εγώ δεν επομίζομαι την ευθύνη των ε, αποτυχιών. Ας πούμε, μπορούμε να πούμε ένας από αυτούς είναι ο Μουγκάμπε. Στη Συρία η αποτυχία είναι ο Ασάντ. Φταίει ο Ασάντ, να το πούμε ξεκάθαρα. Δεν θα συμμετάσχω σε αυτομαστίγωση για να υπομισθώ ευθύνες άλλων. Εν συνεχεία. Να εξετάσουμε και αυτά που ανέφερε ο Κασμάρεκ για την έκθεσή του, τον συγχαίρω, ολιστική προσέγγιση του, Πρέπει όμως να είμαστε άτεγκτοι, υπεύθυνοι για όλες τις αποτυχίες ε, θα πρέπει τελικά να υποστούν τις συνέπειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να τα καταφέρει καλύτερα. Πρέπει να έχουμε καλύτερες αξιολογήσεις στα χέρια μας. Να κάνουμε μια επαναεξέταση πριν καθορίσουμε λεπτομερέστερα τις διεκδικήσεις μας. Merci beaucoup, Monsieur Deva. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Ντέβα. Uh, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Συγχαίρω τον κύριο Κασμάρη και την έκθεσή του. Πληρέστατη. Κάτι που έθιξε ο φίλος μου της Μπέρμαν θέλω να θίξω κι εγώ επιμακρώνει σε αυτή την Επιτροπή και ήταν πολύ καλή η ομιλία που άκουσα μόλις τώρα, με μεγάλο βάθος. Βέβαια, ίσως οφείλεται στη φυσική του ευφυΐα. Αλλά αυτά που είπε, κυρία Πρόεδρε, έχουν σοβαρές συνέπειες για μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατάγομαι από την Ασία και πηγαίνω τακτικά στην Ασία και καμιά φορά βλέπω τη δουλειά μας που παγώνει στο χρόνο. Εμφανιζόμαστε προς τα έξω σαν να μην κατανοούμε τις αλλαγές που γίνονται, τις κοσμοϊστορικές αλλαγές εξουσίες που γίνονται μπροστά στα μάτια μας. Την αλλαγή των αξιών που συνεπιφέρουν οι αλλαγές. Πιστεύουμε ότι διαθέτουμε ευρωπαϊκές αξίες. Και εγώ διάλεξα να μην είμαι πολιτικός στη Σρι Λάνκα, διότι ο θείος μου, ο παππούς μου, ο πατέρας μου, όλοι είχαν αναμειχθεί στην πολιτική ζωή της Σρι Λάνκα. Διάλεξα να κάνω καριέρα κάπου σε μια περιοχή, σε μια χώρα που αισθάνομαι πιο άνετα. Να υπερασπιστώ τις ευρωπαϊκές αξίες που θέλουμε να υπερασπιστούμε. Υποθέτουμε όμως ότι οι αξίες μας είναι παγκόσμιες. Και γι' αυτό συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν σχετικά με την έκθεση Κασμάρεκ. Δεν είναι παγκόσμιε οι καθολικέ και γενικώ αποδεκτέ οι αξίε μα. Είναι ευρωπαϊκέ. δεν θεωρούνται από τι αναδυόμενε δυνάμει Ασία ω τέτοιε παγκόσμιε καθολικέ αξίε επανειλημμένα βλέπω, ιδιαίτερα στην Ασία, παραδοσιακές αρχές από την εποχή της φοδαρχίας. Είναι πολύ παλιά, παλιός πολιτισμός, 2.500 ετών στην Ασία. Και αρχίζουν και κυριαρχούν αυτές οι παλιές αξίες στις καθημερινές δραστηριότητες. Δεν θέλω να αναφέρω μόνο την Κίνα, το Βιετνάμ, στις διάφορες χώρες. Δύο πράγματα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε. Στους νέους στόχους της χιλιετίας θα πρέπει να προβλέπουν την προστασία των ανθρώπων. Θα πρέπει να ελαφρύνουμε, να μειώσουμε την ένδια στο μέτρο του δυνατού. Να έχουν βιώσιμες συνθήκες ε, ζωής στο μέτρο του δυνατού Πρέπει όμω να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε, να προστατεύσουν τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκεί πρέπει να γίνουν μεγαλύτερε προσπάθειε. Και να υπάρξουν σωστέ συνταγματικέ ε, κυβερνήσει. Δεν υποθέτω ούτε στιγμή ότι αυτά είναι δεδομένα. Και όλος ιδιαίτερος η Επιτροπή μας θέλει να ενστερνιστεί αυτές τις πτυχές και να τη στηρίξουμε πιο ένθερμα από ό,τι μέχρι τώρα, κυρίως μέσω του στόχου, του αναπτυξιακού τη χιλιετία. Μέχρι τώρα στην Υποπιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων έχουμε αφήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο, η Επιτροπή μα και οι αναπτυξιακοί στόχοι τη χιλιετία πρέπει να λάβουν υπόψη αυτέ τι αξίε και να είναι ο κινητήρα για την αναπτυξιακή διαδικασία αυτέ οι αξίε. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Κόρτες Λάστρα. Είναι ο τελευταίος που ζήτησε το λόγο στη συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχικά να εκφράσω την πλήρη μου υποστήριξη στα λόγια του συναδέλφου Κάσμαν. Να ευχαριστήσω επίσης και τον εισηγητή για το κείμενο που μας παρουσίασε. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ καθοριστική στιγμή για την μελλοντική πολιτική, την αναπτυξιακή που θα έχουμε. Πολλά ζητήματα ταυτόχρονα έχουν τεθεί, τους στόχους ε, για τις αναπτυξιακές στόχους μετά το 2015, έχουμε την αναθεώρηση το ορισμού της επίσημης αναπτυξικής βοήθειας, έχουμε τη συζήτηση για τη νέα συνολική ε, θεώρηση, τον ρόλο της ε, ασφάλειας και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα συστήματα τα οποία συζητούμε θα μπορούσαν να επηρεάσουν στο μέλλον τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη φτώχεια από το αναπτυξιακό πρίσμα. Ε, και επίσης ε, πώς θα συνεχίσουμε μια επιτυχημένη διαδικασία, κατ' εμέ τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά τους στόχους του αναπτυξιακού χιλιετίας, να πω κάποια πράγματα, τα πιο πολλά τα είπατε. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που έχετε πει, αλλά κάποια είναι σημαντικά. Πρώτα απ' όλα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε στον τομέα, στο, μονοπάτι της εκρίζωσης της στόχης και της ανάπτυξης, αν δεν λάβουμε υπόψη μας τη διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό νομίζω ότι είναι θεμελιώδες και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό. Δεύτερον, δεν θα είναι δυνατόν να εκπονήσουμε ένα νέο γενικό πλαίσιο για την ανάπτυξη σε ένα σενάριο μετά το 2015, εάν, όπως έλεγε ο κύριος Γκέρνς, δεν καταφέρουμε να προβούμε σε μια σε αξιολόγηση το τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, για να αντλήσουμε διδάγματα και να προσδιορίσουμε τις αποτυχίες μας, πώς και γιατί αποτύχαμε. Τρίτον, η όλη συζήτηση, ο προβληματισμός μας για τους στόχους, αναψυχικούς στόχους χιλιετής μετά το 2015, μια συζήτηση που ξεκινάει, θα πρέπει, γιατί τέλος θα αποτύχει, να είναι στο δυνατόν πιο συμμετοχική. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Εθνικά Κοινοβούλια, Περιφερειακά Κοινοβούλια Κοινωνικών των Πολιτών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι μια διαδικασία όπου η, κοινωνική, η κοινωνία των πολιτών που θα παρεμβαίνει θα είναι και αυτή από τι βόρειε χώρε και από το βόρειο και από τον νότο. Και συμμετοχική διαδικασία πρέπει να υπάρχει και να υπάρχει και νομιμοποίηση για να μπορέσουν αυτοί οι στόχοι του 2015 να είναι αποτελεσματικοί τέλο. Κάτι θέλω να υπογραμμίσω και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η διαδικασία στο πλαίσιο των στόχων bla, μέχρι το 2015. Θα πρέπει να έχουμε ένα θεματολόγιο χρηματοδότησης που θα είναι προβλέψιμο και ρεαλιστικό. Αυτή είναι η στόχη που θα καθορίσουμε και που θα πρέπει σε αυτό και το οικονομικό θεματολόγιο, δηλαδή τι ε, προβλέψει τη χρηματοδότηση, να μπορούμε να του εντάξουμε αυτού του στόχου. Αλλιώ δεν θα, έχουμε, δεν θα έχουν, έρθουν σε αίσιο πέρα οι όλε αυτέ οι εργασίε. Θέλουμε λοιπόν και το οικονομικό θεματολόγιο, την οικονομική ατζέντα, να διδαχθούμε από το παρελθόν. Τη βιώσιμη ανάπτυξη, παραλαμβάνω, να την έχουμε ω επίκεντρο για να συζητήσουμε το μέλλον της αναπτυξιακής συνεργασίας που πρέπει να την επαναπροσανατολίσουμε γιατί δεν είναι και στις καλύτερες της εποχές. Ο κύριος Μπέρμαν, να απαντήσω σε αυτά που είπε ο κύριος Ντέβα. Τα λέω γαλλικά, ότως ώστε οι μελλοντικοί ευρωβουλευτές από το Μιγάντ να με καταλάβουν όταν λες ότι οι καθολικές αυτές τις αξίες δεν είναι παγκόσμιες αξίες. Αντιδρώ κάπως. Λέω βέβαια υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές, πολύ μεγάλες καμιά φορά. Όταν μου λες κάτι τέτοιο, πάντα τη σκέφτομαι εκείνον που δεν έχει δικαιώματα, το οποίο τα δικαιώματα παραβιάζονται. Ο Γιωργός στην Αιθιοπία, που δεν μπορεί να πάρει λείπασμα διότι να ανήκει στο κόμμα της εξουσίας. Και ισχύει αυτό. Είναι έλλειψη δημοκρατία που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Και αυτή η έλλειψη δημοκρατία οδηγεί η ανάπτυξη αυτή τη χώρα να αποτελματώνεται πολιτικώ. Εκείνοι που φέρουν από βασανιστήρια. Εκείνοι που είναι αντικείμενα διάκριση. Ε, στην Ουγγάντα, Ε, Κάποιε κάστε στην Ινδία κλπ. Και ελπίζουν μόνο στι καθολικέ αυτέ αξίε αυτοί οι άνθρωποι. Η γυναίκα στη Σαουδική Αραβία. Οι ομοφιλόφιλη στη Σαουδική Αραβία. Σκέφτομαι τα θύματα της έλλειψης, στέρησης δικαιωμάτων. Ε, για όλους αυτούς υπάρχει μια ελπίδα ότι πολιτικοί όπως εσύ, όπως εγώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σηκωθούν και θα πούν υπάρχουν αυτές οι καθολικές αξίες και υπάρχουν για όλους και μετά ε, οι, αυτοί που έχουν την εξουσία λένε μπορούμε να τις σχετικοποιήσουμε αυτές τις αξίες. Γιατί, διότι αυτοί από την έλλειψη δικαίου και δικαιοσύνης ε, υποφελούνται. Δεν το συζητάμε. Ήθελα να προσθέσω αυτά που είπα τώρα σε αυτά που μας είπες. Μία μικρή απάντηση από πλευρά του κυρίου Ντέβα τώρα. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι συμφωνούμε. Αυτό προσπαθώ να πω είναι ότι αυτές οι αξίες που θεωρούμε ότι είναι παγκόσμιες εμβελία καθολική, έχουμε την τάση να υποθέτουμε ότι όλοι τις καταλαβαίνουν και όλοι, τις, ε, ε, όλοι έχουν τις ίδιες αξίες στο σύστημά τους. Δεν γίνεται αυτό και πρέπει να καταβάλουμε παραπάνω προσπάθεια την οποία δεν καταβάλουμε. Δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στον κύριο Γκασπάρ Φραντίνη δίνω το λόγο. Thank you, Ευχαριστώ. Καταρχάς, να καλωσορίσω το σχέδιο έκθεσης που παρουσιάστηκε. Επίσης, να ευχαριστήσω όσους αναφέρθηκαν στην ανακοίνωση της Κομισιόν που υιοθετήθηκε το Φλεβάρι και που την καλωσόρισαν. Νομίζω ότι συμφωνώ με την γενική άποψη της, ε, που παρουσιάζεται στην έκθεση και με τις συστάσεις της. Καλωσορίζουμε κυρίως το γεγονός ότι αυτή η έκθεση λαμβάνει υπόψη της πολλά από τα θέματα και τις συστάσεις που προσπαθήσαμε και εμείς να αναπτύξουμε στην ε, δική μας την ανακοίνωση, οπότε αυτό είναι πολύ θετικό. Νομίζω ότι ε, είναι μια σύγκληση αυτή, σύγκληση απόψεων μεταξύ των όσων κάνουμε στην Κομισιόν και των όσων περιλαμβάνει αυτή η έκθεση από μια άλλη οπτική γωνία. Αν μου επιτρέπετε να αναφερθώ σε κάποια θέματα πάνω στα οποία νομίζω ότι συμφωνούμε για τούτη την έκθεση. Καταρχάς, όπως λέει η έκθεση, πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις και να σκεφτούμε τη νέα πραγματικότητα. Αναφέρεται εδώ, ε, υπάρχουν ε, αναδυόμενες οικονομίες, έχει αλλάξει το ε, τοπίο της οικονομίας της παγκόσμιας, Υπάρχουν θέματα οικονομικής κρίσης, υπάρχουν θέματα βιωσιμότητας, ε, ε, κλιματολογικών αλλαγών. Όλα αυτά πρέπει να τα μελετήσουμε. Πρέπει να βασιστούμε και στους στόχους της χιλιετίας, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις καινούριε προκλήσεις που μας περιμένουν. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, όπως λέει και η έκθεση, να αντιμετωπίσουμε τα θέματα ε, ένδυας αλλά και τα θέματα βιωσιμότητας από κοινού. Και βλέπω ότι υπάρχει όλο και περισσότερη συνένεση ως προς αυτό. Επίσης συμφωνούμε με το γεγονός ότι το νέο πλαίσιο θα πρέπει να είναι καθολικό. Θα πρέπει να καλύπτει όλες τις χώρες και να έχει στόχους για όλες τις χώρες. Θεωρούμε ότι το επόμενο πλαίσιο, όπως το κάνει και η έκθεση, θα πρέπει να ε, επικεντρωθεί ε, στην εξάλληψη της ένδυας. Παρ' όλα αυτά πρέπει να ξεπεράσουμε το θέμα αυτό και να δούμε και θέματα τα οποία δεν κάλυψαν οι στόχοι της χιλιετίας, αλλά είναι ουσιώδη για την αντιμετώπιση την, ε, της ένδυας. Για παράδειγμα, να τονίσω τον σημαντικό ρόλο που έχουν να παίξουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, η, η χρηστή διακυβέρνηση, τα θέματα ισότητας, η δημοκρατία, η ειρήνη και η ασφάλεια που αναφέρονται εδώ. Και να ε, διασφαλίσω εδώ ότι ε, αυτό το σημείο είναι πραγματικά κινητήριος δύναμη για όλες τις πολιτικές μας και για την Κομισιόν. Τέλος, να τονίσω τη σύγκληση απόψεων σε ό,τι αφορά το ότι πρέπει να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας, αλλά η χρηματοδότηση για την για την ανάπτυξη ξεπερνά τι δεσμεύσει μας. Αν θέλουμε να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει για το μετά το 2015, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι θα κινητοποιηθούν. Και αυτό περιλαμβάνει και δημόσιους πόρους και ιδιωτικούς πόρους και διεθνώ και στο εσωτερικό. Ε, ας μην ξεχάσουμε τις δεσμεύσεις μας βεβαίως μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο, κυρίως για τις πιο φτωχές χώρες, αλλά πρέπει να κοινοποιήσουμε και όλους τους υπόλοιπους τρόπου τρόπους χρηματοδότησης που έχουμε. Και επίσης, και συμμερίζομαι αυτό που λέει η έκθεση, πρέπει να επιμείνουμε στην ε, σύγκληση της, ε, και στη συνεκτικότητα των πολιτικών για την ανάπτυξη, γιατί αυτό είναι ένα ε, μέσο εφαρμογής, έτσι ώστε να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει για την μετά το 2015 εποχή να τονίσω τρία πράγματα που είναι σημαντικά για μας τελειώνοντας και αναφέρονται και στην έκθεση. Ίσως ε, όχι ε, ενδελεχώς. Καταρχάς να πω ότι είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη την, ε, την συμπεριληπτική και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει να υπάρχουν απαραίτητοι πόροι για να γίνει αυτό και η ανάπτυξη θα πρέπει να είναι καθολική, ισότιμη και βιώσιμη. Να ανοίγει δηλαδή την πόρτα για μια πράσινη οικονομία. Πρέπει να φροντίσουμε όλοι οι τρόποι που ε, έχουμε για να γίνει αυτό θα περιλαμβάνονται στο, ε, στο νέο αυτό πλαίσιο. Ας πούμε, ενέργεια, ιδιωτικός τομέας, εκπαίδευση, βιώσιμη γεωργία, τηλεπικοινωνίες, κουλουπού. Όπως λέει η έκθεση, και όπως είπα και εγώ, το πλαίσιο θα πρέπει με συνεκτικό τρόπο να αντιμετωπίσει θέματα ενδίας και βιωσιμότητας. Νομίζω όμως ότι πρέπει να πάει και λίγο πιο εκεί. Πρέπει να συγχωνεύσει τα δύο υπάρχοντα πλαίσια σε ένα συνεκτικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να έχουμε στον, σε έναν πλανήτη για τους ίδιους τομείς δύο διαφορετικούς στόχους πρέπει να έχουμε μία δέσμη στόχων που θα καλύπτει και τα θέματα ένδυας και τα θέματα βιωσιμότητας. Πρέπει λοιπόν να περάσουμε μία από μία διαδικασία που θα συνδυάσει, που θα συγχωνεύσει το πλαίσιο ε, για τους, ε, με τους ε, στόχους της χιλιετίας και το πλαίσιο μετά του στόχου τη χιλιετία και θα τα μετατρέψει σε ένα κοινό πλαίσιο και για τα δύο. Αυτή λοιπόν είναι μια διεθνή ε, διαδικασία στην οποία πρέπει να εμπλακούμε. Αυτό ε, το πλαίσιο και αυτοί οι στόχοι δεν θα αποφασιστούν εδώ ούτε μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα θέμα διεθνού εμβέλεια. Είναι μια διαπραγμάτευση που θα γίνει σε διεθνέ επίπεδο και αυτή η διαδικασία θα αποφασίσει τους στόχους. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε έτοιμοι και συντονισμένοι και σε γρήγορση για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε αυτή τη διαδικασία. Και γι' αυτό το πιο σημαντικό είναι να έχουμε σαφή στοχοθέτηση για στα, σαφή προσανατολισμό ώστε να καθοδηγήσουμε σωστά την όλη διαδικασία που θα ακολουθήσει. Χρειαζόμαστε λοιπόν σαφής, ε, σαφή στρατηγική και σαφή διαδικασία. Όλοι μας, και το Κοινοβουλίο και τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν, έτσι ώστε να μπορέσουμε συνολικά να ε, επηρεάσουμε αυτή την ε, διεθνή διαδικασία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος... Κύριε Μαρτίνεθ, έχετε το λόγο. Σας είδα, συγγνώμη. Έχετε το λόγο. Και... Me, hubiera, hubiera, quizá hubiera deseado hablar antes de... Ίσως ε, θα ήταν ε, καλύτερα να είχα μιλήσει πριν από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, αλλά τέλος πάντων δεν θα ε, αντισταθώ στον πειρασμό να μιλήσω για κανένα δύο λεπτάκια. Σήμερα είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική ακρόαση το πρωί. Πάρα πολύ σημαντική. Ναι. Και πρέπει να ξαναευχαριστήσω την Πρόεδρο για την πρωτοβουλία της εξαγωγής της. Αυτό που συζητάμε σήμερα για το μέλλον δηλαδή, πρέπει οπωσδήποτε να λάβει υπόψη θεμελιώδη ζητήματα που είναι και αντικείμενο της δικής μας Επιτροπής. Πώς θα ε, συζητήσουμε για το μέλλον αν δεν έχουμε επίγνωση αυτών που συζητήσαμε σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί γιατί μιλήσαμε. Μιλήσαμε για διαφθορά. Μιλήσαμε για τη διαφθορά που πραγματικά υποσκάπτει ε, και καταστρέφει τις αρψόμενες χώρες. Και την ψυχική συνεργασία υπονομεύει η διαφθορά. Στο σύντροφο, στον φίλο Κατσμάρεκ, πρέπει να μεταφέρουμε τις ανησυχίες μας. Ό,τι κάνουμε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, εάν δεν ελέγξουμε τη διαφθορά, δεν θα έχει καμία ναι. αξία. Θα είναι εντελώς άχρηστο. Το μόνο που θα κάνει θα είναι να συνεχίσει να τροφοδοτεί τη διαφθορά και μια κατάσταση που έχουμε αναπτυγμένες χώρες και αναπτυσσόμενες χώρες. Δηλαδή η αναπτυξιακή συνεργασία, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ως στόχο έχει να πάψουν να υπάρχουν αναπτυσσόμενες χώρες. Σας παρακαλώ, σας ερωτώ, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Λουί που είστε ο εμπειρογνώμων και σας ερωτώ πόσες από τις αναπτυσσόμενες χώρες πόσες από αυτές με τις οποίες συνεργάζεται εντατικά η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 20 χρόνια πόσες από αυτές τις χώρες έπαψαν να είναι αναπτυσσόμενες. Αν ούτε μία δεν έχει πάψει να είναι αναπτυσσόμενη, σημαίνει ότι έχουμε αποτύχει παταγωδός. Και σήμερα μας εξήγησαν στην ακρόση γιατί αποτυγχάνουμε. Και μας το εξήγησαν εμπειρότατοι εμπειρογνώμονες. Και μας τα είπε και η Διευθύντρια Καταπολέμησης ε, της Απάτης. Διευθύντρια της Όλαφ μας τα είπε μας τα είπε κάποιος τυχαίος. Δεν θα παραλάβουμε όλα αυτά που είπαμε το πρωί, κυρίως γιατί πολλοί που είμαστε εδώ τώρα είμαστε και το πρωί. Αλλά στον Κατσμάρεκ πρέπει να του πούμε ότι στην έκθεσή του πρέπει να δώσει έμφαση στο ότι η διαφθορά είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά αποτρέπει τις αναπτυσσόμενες χώρες από το να πάψουν να είναι αναπτυσσόμενες και τελικά αυτό καταστρέφει και την αναπτυξιακή συνεργασία γιατί κάθε φορά είναι περισσότεροι οι πολίτες των χωρών μας που γνωρίζοντας πώς λειτουργεί η αναπτυξιακή συνεργασία έχουν πάρα πολύ ε, θεμητές, δικαιολογημένες αμφιβολίες και ερωτηματοκά για το κατά πόσο θα πρέπει και αυτοί να συνεχίσουν να συνεισφέρουν με τους δικούς τους πόρους αν πάνω στο γκάλαθο των αχρήστων, αν είναι μια τρύπα στο νερό όλα αυτά τα χρήματα. Είδαμε τι έγινε στο Αφγανιστάν. Με κονδύλια που είχαν μπει στη χώρα για την ανισυγκρότηση της χώρας. Ένας πολίτης που δίνει ε, τα δικά του χρήματα, που είναι και λίγα, πάρα πολύ λίγα, και που νομίζω ότι συνεισφέρει στην ανοικοδόμηση, ανασυγκρότηση του Αφγανιστάν, δεν θα εξοργιστεί αυτός ο άνθρωπος όταν λάβει συγκεκριμένες πληροφορίε ότι 900 εκατομμύρια δολάρια συγκεκριμένα εξαφανίστηκαν. Δεν περάσανε, δεν πήγανε όμως, ε, δεν έγιναν ατμός, μπήκαν στις τσέπες κάποιων ανθρώπων. Αν δεν είμαστε σε θέση αυτό το πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε, και σε βάθος μάλιστα όλα όσα κάνουμε θα είναι ουσιαστικά ψαντινολογίες, ενδιαφέρουσες ε, συζητήσεις, ε, αερολογίες όμως επί της ουσίας. Εμείς εδώ έχουμε ευθύνη ως ευρωβουλευτές και πρέπει να την αναλάβουμε αυτή την ευθύνη. Άρα αυτό που έγινε το πρωί να το εκμεταλλευτούμε για να βελτιώσουμε και την δουλειά που έχουμε να κάνουμε το απόγευμα. Αυτά και στο κατανόηση για την παρέμβαση κυρία Πρόεδρε. Μα Μας τελειώνει ο χρόνος, αλλά είναι σημαντικό το θέμα και αυτό. Περιοριστείτε παρακαλώ σε ένα δίλεπτο. Ντέβα Γκέρενς. Ο κύριος Μαρτίνες όντως λέει κάτι πολύ σημαντικό. Και ε, θα συμφωνήσω. Τα τελευταία 40 χρόνια έχουμε δαπανίσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη. Και μετά βλέπουμε κάποια άλλα σημεία του κόσμου, όπως η Κίνα, ας πούμε. Η Κίνα έχει περίπου έχει καταφέρει να περίπου 500 με 600 εκατομμύρια πολιτών της να μην ζουν πια στη φτώχεια. Μάλιστα έχει ξεπεράσει τη ΣΥΠΑ. Αναφέρθηκε σε μια έρευνα την προηγούμενο μήνα. Η Κίνα τώρα με, σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς, έχει γίνει η πιο α, πλούσια χώρα του κόσμου. Έχει απελευθερώσει από την ένδια 500 εκατομμύρια κόσμου. Μιλούμε για ευρωπαϊκές αξίες. Είναι σημαντικό αυτό. Η Κίνα δεν έχει ευρωπαϊκές αξίες. Αν υπάρχει ένα κράτος που είναι α, διεφαρμένο, αυτό είναι η Κίνα. Δεν υπάρχουν ευρωπαϊκέ αξίε στην Κίνα, αλλά κατάφερε να βγάλει όλα αυτά τα άτομα από την ένδια. Το ερώτημα λοιπόν πρέπει να θέσουμε εμεί στην Ευρώπη είναι αν προσπαθούμε όντω να βγάλουμε του πολίτε μα από την ένδια μόνο ή αν χρησιμοποιούμε τις αξίες μας για να το κάνουμε αυτό. Και το πιο σημαντικό είναι οι αξίες μας μπορούν να βοηθήσουν του ανθρώπου να βγουν από τη φτώχεια. Η απάντηση είναι ναι, απαντάει ο κύριο Κάσμαν χωρί μικρόφωνο. Ο κύριο Αρλάκη για δύο λεπτά. Ε, I'm sorry, I didn't follow all this. Λοιπόν. συγγνώμη, δεν παρακολουθήσω όλη τη συζήτηση, αλλά άκουσα κάποια νούμερα, κάποια αριθμητικά στοιχεία για το Αφγανιστάν και για την διαφθορά. Και επειδή μελετήσαμε εις βάθος το θέμα αυτό, κατά τη διάρκεια της ε, εκπόνησης της έκθεσης για το Αφγανιστάν, θα ήθελα να διορθώσω κάποια, κάποια στερεότυπα που υπάρχουν για το Αφγανιστάν και για τη διαφθορά. Είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο, ε, η Ένωση και τα κράτη-μέλη στέλνουν ένα δις ευρώ στο Αφγανιστάν. Ο υπολογισμό που κάναμε εμείς για όλη την βοήθεια στο Αφγανιστάν είναι ότι μόνο 20% των αριθμητικών στοιχείων ε, που υπάρχουν για τη διεθνή βοήθεια στο Αφγανιστάν φτάνουν στους Αφγανούς πολίτες. Αλλά προσέξτε, 80% αυτών των κονδυλίων δεν πάει σε αφγανικά χέρια καθόλου. Είναι τεράστιο το λάθος που υπάρχει και είναι ευρέως δεδομένο. Γιατί? Οι περισσότεροι από το μεγαλύτερο κομμάτι της βοήθειας, δηλαδή πάνω από 70% της βοήθειας, δεν περνάει από αφγανικά διάβλους. Μόνο το 30% ή και λιγότερο της βοήθειας περνάει από, ε, ε, από διάβλους. Οπότε εδώ είναι, ο δρόμος, εδώ είναι το σημείο για να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά, όχι στο Αφγανιστάν. Ακόμη και αν πάνω από 50% της βοήθειας που διαχειρίζεται η ε, αφγανική κυβέρνηση περνάει από διάβλους διαφοράς, εξακολουθείτε να έχετε ένα μεγάλο ποσό το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την αφγανική κυβέρνηση ή τον αφγανικό λαό. Οπότε ε, χρησιμοποιήστε προσεκτικά τα αριθμητικά στοιχεία. Το θέμα είναι το πώς φτάνει η τον αυγανικο λαο οποτε χρησιμοποιηστε προσεκτικα τα αριθμητικα στοιχεια το θεμα ειναι το πως φτανει η βοηθεια στους ε, πολίτες. Δαπανάτε, ε, σπαταλιέτε Δεν είναι εκεί λοιπόν μόνο ο τρόπος για να λύσουμε το θέμα της διαφοράς. Είναι και εδώ. Ευχαριστώ. Ο αριθμός των 900 εκατομμυρίων που αναφέρθηκε προέρχεται από μια συζήτηση που είχαμε χτες όσον αφορά την τράπεζα της Καμπούλ, Καμπούλ Μπάνκ, όπου τίθεται θέμα του ποσού των 900 εκατομμυρίων. Και είναι κάτι που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα. Και δεν φταίει σε τίποτα αυτή την απώλεια. Ο κ. Γκέγαν. Λυπάμαι ότι ξεπετάμε στα γρήγορα το θέμα της στρατηγικής και της τακτικής που θα ακολουθήσουμε στις διαπραγματεύσεις. Υποθέτω, και δεν είμαι μόνος που θα το κάνει αυτό, ότι ο Πίμπαλξ θα, θα είναι ο πρώτος στο χώρο. Δεν είμαι σίγουρος ποιος θα τοποθετηθεί, ποιος θα μιλήσει εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε αυτή τη διάσκεψη της Νέας Υόρκης. Γίνονται προσπάθειες για να υπάρξει συντονισμός των θέσεων των κρατών μελών. Θα ήθελα να ξέρω αν οι νέες διατάξεις της συνθήκη της Σαβώνας καλούν και τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθούν. Εμείς πρέπει να επαγρυπνούμε σε αυτό το θέμα και να φροντίσουμε η Ευρώπη να μην παρουσιάζεται κατακαιρματισμένη, αλλά σαν αποφασιστικός φορέας που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Εγώ θα ήθελα να ξέρω, θα ήθελα να ξέρω ποιος θα μιλήσει εκεί. Ποια θα, ποιος θα είναι ο ρόλος μας, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις ενδεχομένως θα πρέπει να προβλεφθεί μια συνεδρίαση με τον ή τους υπευθύνους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θα πάνε στη Νέα Υόρκη να παρουσιάσουν τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν γίνεται αλλιώ, ίσω μπορεί να ετοιμαστεί και κλεισμό των θηρών συνεδρίων των συντονιστών. Διότι το θέμα τη στρατηγική και τη τακτική, αυτά τα θέματα, δεν συζητούνται δημοσία. Σημειώνουμε δεόντως το αίτημα του κυρίου Γκέρεντς να συντονιστούμε πριν τη Νέα Υόρκη το φθινόπωρο. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ζήτησε το λόγο. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μίτσελ για να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση σχετικά με τους νέους αναπτυξιακούς στόχους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που επιτρέπετε στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης να προβεί σε κάποια σχόλια και να συμπληρώσει τα όσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ανακοίνωση με τίτλο «Αξιοπρεπή ζωή για όλους» είναι πολύ σημαντική. Και για μας. Εμπλεκόμεθα και εμείς στην επεξεργασία της. Και η κυρία Κάθια Στον συμμετείχε στην όλη προσπάθεια. Είπατε εκπρόσωπος. Κάποιοι αναφέρθηκαν στην ανάγκη να μάθουμε από το παρελθόν τι λειτουργήσε, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά όσον αφορά από το πλαίσιο των στόχων της χιλιετίας. Να αναφέρω, κάποια στοιχεία ε, της ανακοίνωσης που προέρχονται από τα μαθήματα που αντλήσαμε από το εγχείρημα και που τα υποστηρίζει η υπηρεσία μας. Ποια είναι τα στοιχεία λοιπόν. Πρώτα απ' όλα ισότητα, ισοτιμία, δικαιοσύνη. Από την άλλη πλευρά ασφάλεια, ειρήνη. Η ανακοίνωση προβάλλει τη σημασία αντιμετωπίσεως αυτών των θεμάτων την περίοδο μετά το 2015. Διότι είδαμε ότι υπήρξαν κάποιες ε, αδυναμίες όσον αφορά την προσπάθεια κρίζωσης της ένδυας. Και γι' αυτό διηγηθήκαμε σε κάποιες αποτυχίες ή σε μερική επιτυχία. Η δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι μόνο κρίσιμα για την πρόοδο, για την ανάπτυξη, αλλά και σημαντικότατες αξίες, αυτές καθεαυτές. Το ίδιο ισχύει για την ειρήνη και την ασφάλεια. Είδαμε ότι ελάχιστη πρόοδος, σχεδόν μηδενική, σε εύθραυστες χώρες σε περίοδο μετά από συγκρούσεις. Οπότε οποιοδήποτε πλαίσιο καθοριστεί για μετά το 2015 θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και αυτά τα ζητήματα. Με τα χαράς βλέπουμε ότι αυτά τα δύο θέματα καλύπτονται στο σχέδιο εκθέσεως του Κοινοβουλίου. Και θα θέλαμε να παραμείνουν και να ενισχυθούν περαιτέρω. Ευχαριστώ. Κύριε Μίτσελ, σας δίνω το λόγο για να ολοκληρώσετε. Ναι, μπορώ να είμαι πάρα πολύ σύντομος, κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα όλους όσους έλαβαν το λόγο. Είναι εδώ η συνεργάτη του κύριου Κάτσμαρ και θα σημειώσω όλα τα σχόλια. Τέσσερα, ε, έτσι, πολύ τηλεγραφικά ως απάντηση σε σχέση με αυτά που είπε ο Σάρλ. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο συντονισμός, θα πρέπει να το συζητήσουμε και σε επίπεδο συντονιστών με το Συμβούλιο και τον Επίτροπο Πίμπαλξ. Θα πρέπει να υιοθετήσουμε με μια ενοποιημένη, μια ενιαία προσέγγιση για αυτούς τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα δαπανών ταξίκρατων μελών και ένωσης. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και ελπίζω να ληφθεί υπόψη και στο πλαίσιο μετά το 2015. Η διεθνή κοινότητα ε, πρέπει αυτό το ζήτημα να το συζητήσει. Γιατί έχουμε τέτοια έλλειψη αποτελεσματικότητας. Επανέρχομαι ε, όμως αυτό που είπε ο κύριος Μαρτίνεθ για τη διαφθορά και εφιστώ την προσοχή του κυρίου, θα επιστήσω μάλλον την προσοχή του κυρίου Κατσμάρη στο θέμα αυτό, γιατί συζητήσαμε το πρωί όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα και στο γεύμα συζητήσαμε και τα περί διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα περί ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε τέτοιε ρήτρε ίσω και στι διεθνεί μα συμφωνίε. Ο κύριος Ντάτσκας μίλησε για τη μη χρηματοοικονομική βοήθεια, δηλαδή ε, την μετάδοση γνώσης και τεχνογνωσίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί πόροι στα κράτη-μέλη, ακόμη και μεταξύ των τοπικών αρχών των κρατών μελών. Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι πόροι αυτοί στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αυτό σωστά πρέπει να μας απασχολήσει για το επόμενο, για την αναθεώρηση των στόχων αυτών μετά το 2015. Ευχαριστώ όλους όσους ε, συνεισέφεραν και ελπίζω να υιοθετήσουμε μια συντονισμένη προσέγγιση για τη Νέα Υόρκη αργότερα φέτος. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Alors, il y a un changement Εναλλαγή βλέπω, άλλη ομάδα επισκεπτών ε, μπαίνει στην αίθουσα για να παρακολουθεί τις εργασίες μας. Και θέλω να καλωσορίσω όλους όσους ε, ήρθαν, να σας ε, χαιρετήσω. Είστε από το Μάλμο, από τη Σουηδία. Και ήρθατε να παρακολουθήσετε τις εργασίες της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μιλήσουμε για το Μάλι ε, συγκεκριμένα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στα γαλλικά η Τώρα περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της μέρης διάταξης. Ah ah Συγγνώμη, αλλά ξέχασα να πω ότι η πολύ σημαντική έκθεση του κύριου Κατσμαρέκα μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι το, τις 12 το μεσημέρι 25 Μαρτίου και στις 23 Απριλίου θα ψηφίσουμε. Λοιπόν, τώρα περνάμε στο σημείο 16 της μερισιάς διάταξης, Μαλή. Έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ ένα μέλος επιτροπής που δεν το βλέπουμε και πολύ συχνά, τον κύριο Λίνι ο οποίος είναι συμπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Και υπό την ιδιότητα του, του Προέδρου ε, συμμετείχε σε μια αντιπροσωπεία στο Μαλί πρόσφατα με στόχο να ε, εκτιμηθεί η κατάσταση ε, στη χώρα, σε αυτή την εμπόλεμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Αντιπροσωπεία στο Μαλί λοιπόν ενέκυψε σε μια σειρά ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη, ανοικοδόμηση ε, μάλλον ε, αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών, ηλεκτροδότηση στον Παμάκο για παράδειγμα και όλο ιδιαίτερο υπηρεσίες υγείας, παιδεία, δημιουργία θέσεων απασχόληση. Επίσης, ετέθη το ζήτημα τη προετοιμασία για τη διεξαγωγή εκλογών στη χώρα. Ένα άλλο ζήτημα που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε είναι η σφαιρική συνολική προσέγγιση απέναντι στην κρίση της περιοχής του Σαχέλ. Το Μάρτιο του 2011 την εγκρίναμε στο Κοινοβούλιο και για πρώτη φορά θα δοκιμαστεί η προσέγγιση αυτή στο Μαλί. Βασίζεται σε στενές άμεσες σχέσεις μεταξύ ανάπτυξης και ασφάλειας. Το ένα σκέλος ενισχύει το άλλο και πρέπει να δοθεί μια περιφερειακή απάντηση σε μια πολύπλοκη, πολυσχηδή κρίση. Νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να συζητήσουμε και για τις αλληλεπιδράσεις αυτών των δύο ε, αξώνων, δηλαδή ασφάλειας και ανάπτυξης, για να έχουμε μια συνολική συνεκτική προσέγγιση. Δεν θέλω να με ακρηγορήσω άλλο και θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μας ευθύ αμέσω. Κύριε Λουί Μισελ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν έρχομαι συχνά στην τριάση σας γιατί είμαι ένας ταπεινός αναπληρωτής του συναδέλφου Αλγκέρνας που τα έχει τα θέματα πολύ καλύτερα από εμένα. Όταν είναι αυτός είναι σαν να ήμουν εγώ παρόν. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πράγματι ήμουν επικεφαλής πρόσφατος ε, μιας αντιπροσωπείας μελέτης και ενημέρωση στο Μαλί εξ ονόματος της Ισομερούς ε, της Συνέλευσης Εκπροσώπησης ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Χωρών ΑΚΕ με συνόδευαν ο η Μισελ Ριβαζή και, ο, και η Φρανσουάς Καστέξ, εκλεκτοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας αναφέρω ορισμένες ε, σκέψεις μετά από την ε, αντιπροσωπεία αυτή, μετά την αποστολή αυτή. Συνολικά πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά την κατάσταση πριν τη γαλλική επέμβαση. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι πρόοδος έχει επιτευχθεί και είναι σημαντική. Όμως, η αυτή φυσικά και δεν μπορεί να κρύψει τους κινδύνους που εξακολουθούν να ελοχεύουν. Πρώτον, πρέπει νομίζω να συγχαρούμε τον Γάλλο Πρόεδρο και τη Γαλλική Κυβέρνηση τον Φρασό Αλόντ λοιπόν και τη γαλλική κυβέρνηση πρέπει να ε, πούμε ότι ε, αξίζουν πολύ μεγαλύτερη ε, υποστήριξη και εκτιμήσεις, διότι άλλαξε τα δεδομένα ριζικά και δεν είναι απλό αυτό. Μπορεί κάποιες ευρωπαϊκές χώρες να κινητοποιήθηκαν, μένα, αλλά πρέπει να πούμε ότι το έκαναν ε, έτσι πολύ ε, με το ζόρι, θα έλεγα, και ήταν κατώτερη των προσδοκιών σε μια τέτοια κατάσταση η συμμετοχή τους. Νομίζω ότι πολλές ε, χώρες ευρωπαϊκές παραμένουν στο επίπεδο των ε, ωραίων λόγων, ε, μεγάλα λόγια, αλλά πολύ λίγες οι πράξεις που συνοδεύουν τα λόγια. Πρέπει επίσης να δώσουμε έμφαση στον ενδιαφέροντα ρόλο του Τσάντ. Ο, ο ρόλος του στρατού, των ενόπλων δυνάμεων του Τσάντ δεν ήταν ελάσσον τα κράτη-μέλη δεν ε, συνεισφέρουν επαρκώ αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε. Η ανάλυση μα λοιπόν μα κάνει να απευθύνουμε έκκληση ώστε η συνεισφορά και σε άνδρες και σε ε, υλικοτεχνική διοικητική μέρημνα και σε εξοπλισμό να είναι στο ύψος των ε, προκλήσεων στο Μαλί. Θέλω να σας πω ότι πηγαίνοντας επί τόπου αντιλαμβάνεται κανείς τον πόλεμο που βλέπει στο βόρειο του Μαλί ότι ο πόλεμο αυτός ξεπερνάει το Μαλί. Μπορεί κάποιο να έχει την εντύπωση ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορά μόνο το μαλλί. Όχι, όλου μα μας αφορά και πάρα πολύ άμεσα. Αφορά βέβαια και το μαλλί, αλλά αφορά και την όλη ευρύτερη περιοχή. Αφορά ε, την Αφρική, αφορά την Ευρώπη και αφορά τον κόσμο ολόκληρο. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο συμπέρασμα και νομίζω ότι πρέπει και ίσως ως κοινοβούλιο θα μπορούσαμε να κινητοποιηθούμε. Δεν μπορούμε, τουλάχιστον εγώ είμαι πεπισμένο μετά από την ε, αποστολή αυτή, δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Γαλλία μόνη τη πέραν σε αυτή την πρόκληση. Μας δείχνει κάποιε πραγματικότητες ε, η αντιπροσωπεία αυτή. Πολλές φορές υπάρχει μια καταπροσέγγιση ε, εντύπωση της πραγματικότητας και ε, αυτό καταρρύπτεται από τα απορίσματα αυτής της αντιπροσωπής. Πρώτα απ' όλα, όπως και είπα, ε, δεν είναι μια ε, σύγκρουση εθνική που έχει να κάνει με τους του ή με το ε, αλλά έχουμε πάρα πολλές οργανώσεις που ουσιαστικά ήταν κάποια εξωτερικά μεν, εξωτερικοί παράγοντες που κινήματα ε, τα οποία επηρέασαν την κατάσταση και επειδή έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα, τσιχαντιστές ε, που τηρούν τα νήματα, η τρομοκρατία είναι μια παγκόσμια απειλή. Ε, στην Ιναμένα, στην Αλγερία είδατε τι έγινε με την τρομοκρατική απόπειρα εκεί. Άλλη, άλλο συμπέρασμα. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε και γι' αυτό δεν γίνεται συχνά λόγος κατά την άποψή μου, αλλά παραμένει μια απειλή. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τη θέση και το καθεστώς ε, του Σανόκου. Γιατί δεν γίνεται λόγος πολύ γι' αυτόν, αλλά είναι πλέον πρόεδρος της Επιτροπής ε, για τη μεταρρύθμιση της ασφάλειας. Παραμένει όμως ε, ανησυχητική η προσωπικότητα αυτή για μένα. Έχει πάρει με πολύ μεγάλη ελαφρότητα αυτά τα νέα καθήκοντα και νομίζω ότι θα μπορεί πραγματικά να επηρεάσει πολύ περισσότερο τα πράγματα. ξέρετε τι κάνει, πηγαίνει από τη μια ιεραρχία στην άλλη, ουσιαστικά είναι σαν ένας συνδικαλιστής, ένα φερέφωνο των διεκδικήσεων των στρατιωτικών. Έχει δηλαδή ε, την πλήρη προσοχή των ε, στρατιωτικών. Και παίρνει και ένα προεδρικό μισθό γιατί το διαπραγματεύτηκε αυτό. Ο λόγο κύριος δηλαδή ζει μέσα σε μεγάλες ανέσεις. Αυτό που νομίζω ε, είναι ότι δεν πρέπει να υποτιμήσουμε σε καμία περίπτωση τον καταστροφικό ρόλο που θα μπορούσε να παίξει. Είναι σε θέση και ίσως είναι ο μόνος σήμερα και παρά τη γαλλική παρουσία να δημιουργήσει πραξικόπημα, να προκαλέσει πραξικόπημα, γιατί τη, κινεί τα νήματα στο στρατό. Και αυτό είναι ανησυχητικό για μένα. Και πρέπει να το πούμε. Επόμενο. Πριν μιλάμε για το στρατό, Η διεθνή εταίροι νομίζω ότι πρέπει να επιταχύνουν και όταν επιταχύνουν, να επιταχύνουν τάχιστα την αναδιάρθρωση του στρατού. Εκπαίδευση επιμόρφωση. Δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την αποστολή. Και πρέπει να το συνεχίσουμε ε, το εγχείρημα αυτό και να το στηρίξουμε ακόμη περισσότερο. Μια ακόμη πεποίθησή μου μετασχηματισμό τέλο πάντων μεταφορά τη μίσμα τη διεθνού δηλαδή αποστολή υποστήριξη στο Μάλι. Υπό αφρικανική ε, διεύθυνση. πρέπει να κάνει peacemaking ε, αυτή η αποστολή. Υπάρχει αυτή η διαφορά peacemaking, peacekeeping. Τεράστια η διαφορά. Εδώ έχουμε συζήτηση όχι για peacemaking αλλά για peacekeeping. keeping όμως πρέπει να λάβουμε τις ευθύνες μας ως κοινοβούλιο σε σχέση με αυτό. Και πρέπει να ασκήσουμε peace. Να μην είναι απλά peacekeeping, αλλά να είναι και peacemaking. Και θα πρέπει και τα στρατεύματα του ΟΗΕ που είναι εκεί να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, την ισχύ τους. Να μην έχουν μόνο μια διαχειριστική ε, στάση, να μην είναι παθητική. Πρέπει να μπορούν να ε, δράσουν. Άρα πρέπει να έχουν και μια πραγματική εντολή άρθρο 7 ενισχυμένου. Μιλάμε για διατήρηση της ειρήνης ε, υπ' αυτή την έννοια, αλλά ε, αυτό προκαλεί κάποια παρανόηση ε, στους κατοίκους. ότι αν κάνουμε peacekeeping τελικά, κατά κάποιο τρόπο, καθιερώνουμε αυτό το διχασμό, αυτή τη διχοτόμηση. Θέλουμε να διαχωρίσουμε ε, τις ε, εμπόλεμες πλευρές. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτό το επιχείρημα, που είναι πολύ πιστικό. Τέταρτη πεποίθηση. Το είπε και ο Γάλλος Υπουργό Άμυνα πριν από κάποιε μέρε. Πρέπει το στομότερο δυνατόν, και το πιστεύω και εγώ, να ξεκινήσει πολιτική διαδικασία. Έχει πολύ δίκιο ο Γάλλος Υπουργό Άμυνα. Η διαδικασία αυτή νομίζω πρέπει να βασίζεται σε τρει απαιτήσει. Υπάρχει τεράστια συζήτηση γύρω από όλα αυτά, αλλά εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένο ότι πρέπει πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, να οργανωθούν εκλογές για να ε, σταματήσει αυτή η μεταβατική φάση. Καλό είναι το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης. Προτείνουν την 7η Ιουλίου για τον πρώτο γύρο, 30 Ιουλίου για το δεύτερο. Ο Ιούλιος μου φαίνεται ότι είναι μια ε, πιθανή, μια δυνατή ημερομηνία. Ο υπουργό ε, ε, για τα διοικητικά θα είναι τη εκλογές τον συνάντησα, αλλά συναντήθηκε με τον πρόεδρο τραρέ, με τον πρωθυπουργό, με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου τη Συνέλευσης, τον κύριο Κολυμπαλή, τον συνάντησα και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Συναντήσαμε και βουλευτέ από το Βορρά, την κοινότητα των πολιτών από το Βορρά τη συναντήσαμε. Είχαμε καλέσει επίση. εκπροσώπου από θρησκευτικέ οργανώσεις, καθολικοί ήρθανε, Κάποια άλλα δεν αποκρίθηκαν, τέλο πάντων. Λίγο πολύ συναντήσαμε όλου. Υπάρχει μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει. Το θέμα είναι αν είναι το timing τέτοιο ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε εκλογέ στον Ιούλιο, στο Μάλι. Η πρόεδρο μπορεί να ρυθμίσει ε, το πρόβλημα το οποίο παραμένει. Ποιο είναι αυτό. Οι βασικέ υπηρεσίε σήμερα, μάλλον το, το ανέφερε, οι βασικέ υπηρεσίε σήμερα δεν έχουν αποκατασταθεί διοικητικές υπηρεσίες. Δεν έχουν δρομολογηθεί πάλι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έφυγαν, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την επαναποκέντρωση και υπάρχουν και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπιστέντες ή πρόσφυγες. Δηλαδή είτε εσωτερικά εκτοπιστέντες είτε εξωτερικά, άρα πρόσφυγες. Και είναι μια σημαντική εκλογική μάζα. Μπορεί να είναι 500.000 με τον πρόεδρο, με τον κ. Ωρέ, θα συζητήσαμε και ίσως η μόνη υποχώρηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς, ε, η προσωπική μου άποψη μάλλον είναι αυτό, για το timing, είναι σημαντική η άποψη της διεθνούς κοινότητας, είναι να αποσυνδέσουμε τις προεδρικές εκλογές από τις βουλευτικές εκλογές. Γιατί, γιατί οι προεδρικές εκλογές, γιατί έχουμε μία και μόνη εκλογική περιφέρεια, κάτι που δεν ισχύει για τις βουλευτικέ εκλογές, οπότε μπορεί επί επιτόπου ε, να ψηφίσουν και οι εκτοπιστέντες και οι πρόσφυγες. Αυτό εύκολα μπορεί κανείς να το οργανώσει. Άρα μπορούν τον Ιούλιο να γίνουν οι προεδρικές εκλογές. Έτσι θα υπάρξει μια επανανομιμοποίηση ε, μια αρχής. Δεν θα έχουμε δηλαδή πια μετάβαση, μεταβατική περίοδο. Και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα αντίποδα σε απόπειρε πραξικοπήματο. Και μετά τον Οκτώβριο να οργανωθούν βουλευτικέ εκλογέ. Είναι ένα χρονοδιάγραμμα που μα φαίνεται πιθανό, εφικτό. Για τι βουλευτικέ να πω ότι οι βασικέ υπηρεσίε θα πρέπει κατ' ένα ελάχιστο, στοιχειοδό, κατ' ένα ελάχιστο επίπεδο να λειτουργούν. Ούτε τα σχολεία όταν πήγαμε δεν είχαν ξαναλειτουργήσει, Αλλά αυτά θα πρέπει να τα δημιουργήσουμε. Οι δάσκαλοι δεν είναι πλέον στις περιοχές που δίδασκαν και ούτω καθεξής. Αυτό είναι σημαντικό. Να σας πω ότι αυτό που χρειάζεται να εργοποιηθεί η Επιτροπή Διαλόγου και Συμφιλίωσης. Εκεί κάποιες δυνάμεις μπορούν να χειραγωγήσουν τις εκλογές και λένε ότι θα πρέπει πρώτα αυτή η Επιτροπή για το Διάλογο και τη Συμφιλίωση να δώσει τις συστάσεις πριν γίνουν οι εκλογές. Ε, έτσι θα γίνουν εκλογέ πριν 4-5 χρόνια. Για να μπορέσει αυτή η Επιτροπή Διαλόγου και Συμφιλίωσης να παραγάγει τα πορίσματά της πριν τι εκλογέ, θέλει τουλάχιστον δύο χρόνια. Η Επιτροπή Συμφ... Διαλόγου και Συμφιλίωσης ε, θεσπίστηκε όταν ήμασταν εκεί. 33 μέλη, εκπρόσωποι όλων των ρευμάτων, αλλά, πώς να το πω, με μια ευχή που διατυπώσαμε ότι θα πρέπει αυτή η Επιτροπή να οργανώσει και αποκεντρωμένους διαλόγους ούτως ώστε να μπορούν όλοι να συμμετάσχουν στις συζητήσεις. Και η γίνει στη συμμετοχή πρέπει αυτοί που συμμετέχουν να πρέπει να δεσμευτούν να, να σεβαστούν την εδαφική ακεραιότητα και να μην έχουν πλέον όπλα. Το καταλαβαίνω αυτό. Να μην χρησιμοποιούν στρατιωτικά μέσα ή βίες μεθόδους για διεκδικήσεις τους. Τρίτη απέτηση, η περιφερειακή διάσταση. Άκουσα αυτό να ακούγεται, εγώ είμαι πεπισμένος βαθύτατα και άκουσα τη συζήτησή σας για το στόχο της χιλιετίας. Σημερίζομαι κατά πολύ αυτά που υπόθηκαν εδώ. Εγώ πρέπει να πω ότι ένα από τα σφάλματα που διαπράττουμε κυρίως στην Αφρική είναι να κάνουμε διμερή ανάπτυξη. Να μην τονίζουμε επαρκώς την περιφερειακή ανάπτυξη. Νομίζω ότι είναι ένα από τα μεγάλα σφάλματα που διαπράττουμε. Και τα διαπράττει αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι δική δικοί μας κανονισμοί, δικές μας διαδικασίες που ακολουθούμε. Είναι ανοησία. Θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε για ανάπτυξη περιφερειακή, πραγματικά ολοκληρωμένη, παρά να κάνουμε αυτό που κάνουμε διμερείς ε, συμφωνίες συνεχώς. Δεν θα υπάρχει συμφωνία ούτε στο Μαλί, ούτε σε άλλα σε αυτή την περιοχή της Αφρικής αν δεν μπούμε πραγματικά σε μια διάσκεψη πραγματική περιφερειακή συμφωνία. Διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό που είπα. Γιατί λέω ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους φίλους μας τους Γάλλους, διότι πιστεύω ότι ακόμα και αν ρυθμίσουν το πρόβλημα του Μαλή, διότι θα το ρυθμίσουν το πρόβλημα στο Μαλή, διότι θα κάνουν καθαρίσεις, θα καθαρίσουν το Μαλή από όλους τους θύλακες τους εξτρεμιστικούς, ο κίνδυνος είναι τεράστιος το πρόβλημα το κακό να μετακινηθεί και να πάει αλλού στη γειτονιά διότι φορά, μισεί το κενό η φύση. Από τη στιγμή που το πρόβλημα του Μαλή θα ρυθμιστεί στατιωτικά, είναι προφανέ ότι θα πάνε αλλού αυτοί για να κάνουν το κακό του, θα πάνε αλλού να δημιουργήσουν προβλήματα. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται πραγματικά μια περιφερειακή σφαιρική προσέγγιση για να ρυθμιστεί το θέμα αυτό. Ιδού κυρία, θα μπορούσα να μακρηγορήσω περισσότερο, αλλά δεν ήθελα να χρονοτριβήσω περισσότερο, να πάρω το χρόνο σα. Πιστεύω ότι σα έδωσα αρκετά στοιχεία για να σκεφτείτε τα θέματα, να διεξαχθεί συζήτηση. Είμαστε στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την εισαγωγή στη συζήτηση. Κύριε Μπέρμαν, έχετε το λόγο. Merci, Madame la Présidente. En fait, juste pour appuyer l'excellent discours de Louis Michel, il me semble que... Έξοχη παρουσίαση του Louis Michel. Face à la France, je me sens simplement honteux. Ντρεπόμαστε όσον αφορά τη θέση μα εναντί τη Γαλλία διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της κάνουν ε, τα πάντα να μείνει μόνη της η Γαλλία, μόνο ε, λόγια λένε. Και στέλνουμε μόνο τεχνικούς συμβούλους για να, να βοηθήσουν το στρατό του Μαλή. Η Γαλλία λοιπόν μένει μόνη της με τους κινδύνους που αναλαμβάνει. Και κάνουμε σαν να μην υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Λεμόντε έλεγε κενό στην Ευρώπη, ε, έγραφε, με επικρίσεις για την Ευρώπη. Διακυβεύματα ευρωπαϊκά και παγκόσμια αυτά που αντιμετωπίζονται. Υπάρχουν νέοι που εκπαιδεύονται και προσιλητίζονται από τους αλαφίστες, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στην Τινησία, στην Αίγυπτο, για να πάνε να πολεμήσουν στη Συρία. Πώς θέλετε να σταματήσει αυτό, αν δεν σταματήσουμε διαπάντως, διαπαντός αυτή την ύπαρξη της Αλκάιντα και των Σαλαφιστών στο Μαλί και γύρω από το Μαλί. Πώς να σταματήσουν αν δεν συνεχίσουμε και αν δεν υποστηρίξουμε την πολιτική, την αναπτυξιακή και στις χώρες της γειτονίας και στις χώρες του Σαχέλ. Στη χώρα μου, στην Ολλανδία, γίνεται συζήτηση σκανδαλώδης κατά την άποψή μου. Να μειωθεί η αναπτυξιακή βοήθεια. Απομονωτισμός διακηρύσσεται. Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα καταστροφικός απομονωτισμός για τα συμφέροντά μας. Δεν καταλαβαίνουμε τα κράτη-μέλη και τα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά εμεί σέρνουμε τα πόδια μα, αντιστεκόμαστε. Η κυρία Γκρέ, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ίσως εγώ θα μιλήσω πιο ελεύθερα, διότι είμαι Γαλλίδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω βεβαίω τον παρεμβαίνοντα, αλλά να κάνω και κάποια σχόλια, παρατηρήσει, να θέσω και ερωτήσει. Δεν λέω ότι είναι φιλανθρωπική η χώρα μου. Αν η Γαλλία παρενέβη, δεν το έκανε κατά τύχη. Δεν υπάρχει συμφέρον της Γαλλίας να είναι σταθερή η περιοχή. Όταν λέω περιοχή εννοώ ευρύτερα περιοχή. Διότι υπάρχουν πρώτες ύλες στην περιοχή. Το επενθύμησα. Υπάρχει ουράνιο. Από αυτό εξαρτώμαστε απόλυτα για τον πυρηνικό μας τομέα. Και αυτά θα πρέπει να επενθυμιστούν. Δεν πρόκειται περί παρεμβάσεως διότι υπάρχουν Ισλαμιστές εκεί αν δεν είχαμε την ανάγκη των πρώτων αυτών υλών, δεν είμαι σίγουροι ότι θα βιαζόμασταν τόσο πολύ με τον ίδιο τρόπο για να υπερασπιστούμε τη σταθερότητα τη περιοχής. Αυτό είναι μια ερώτηση και άποψη. Μια ερώτηση μετά προς εκείνους, προς τους συναδέλφους που πήγαν στο Μάλι και τις βιοπραγίες που έκαναν αντί των αμάχων τον ΠΟΕΛ και των, ε, του ΑΡΕΚ που έκανε ο στρατός του Μαλή, που όλο και πιο συχνά αναφέρονται. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι πληροφορίες έχετε. Υπερασπιστήκατε κάποιο χρονοδιάγραμμα για τις εκλογές και συζητούνται ήδη τεχνικές λεπτομέρειες των εκλογών. Εγώ δεν είμαι καθόλου ειδική για το Μάλι, το λέω, Ξέρω ότι από το 1990 έγιναν εκλογές ε, με εναλλαγές, υπήρχε δημοκρατία στο Μάλι και πάντα άκουγα ότι είναι πρότυπο δημοκρατίας ε, το Μαλί στην ε, Αφρική. Όμως διαπιστώνουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν ακολούθησε, η φτώχεια παρέμεινε και τέλος αυτή η έλλειψη της ανάπτυξης οδήγησε στην ανάπτυξη εξτρεμιστών και τελικά πραξικοπήματος. Δεν ξέρω. Θέτω ερωτήματα. Δεν έχω τις απαντήσεις τα πάντα. Δεν με κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν νέες εκλογές θα αρκέσουν. Θα νομιμοποιήσουν ενδεχομένω μια νέα αρχή. Το ερώτημα είναι για να κάνει τι. Ε, δεν θα ξαναντιμετωπίσουμε την ίδια κατάσταση μετά. Μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε περισσότερο να δημιουργηθεί μια συνέλευση συντακτική να κάνει απολογισμό της περίοδου, να δει τι λειτουργήσε, τι δεν λειτουργήσε, να προβεί σε μια ανάλυση των οικονομικών πολιτικών, να κάνει μια ανάλυση των δημοσίων πόρων, πώς να χρηματοδοτηθεί η παιδεία, η υγεία, να σχηματίσει ένα σχέδιο και να συγκεράσει όλες τις πολιτικές. Έθεσα τις ερωτήσεις, βέβαια, Έχω πάει σε αποστολέ εκλογικέ και αλλού. Θα τα καταφέρουμε και αυτή τη φορά. Θα είναι καλό να έχουμε νέε εκλογέ. Αν γίνουν οι εκλογέ, δεν θα αντιμετωπίσουμε την παλιά κατάσταση αν δεν επιληθούν τα παλιά προβλήματα, αν δεν τεθούν αυτέ οι ερωτήσει. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Ντεκάιζερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μα ποια είναι τα πραγματικά ζητήματα και ερωτήματα Ποια είναι τα ερωτήματα που πρέπει να θέσουμε, τι λύσεις πρέπει να ζητήσουμε. Αυτό που μπορώ να πω μετά από την παρουσίαση από το Λίνι είναι ότι είναι δύσκολο να μην μιλήσουμε για μετατόπιση των κινδύνων. Εδώ ε, το έθιξες, είπες στην αρχή και μετά ανέφερες ε, τρομοκρατικές ε, οργανώσεις, ισλαμικές και άλλες βλέπουμε ανάφληξη της Λιβύης και αυτό είναι το θέμα. Δεν λέω ότι δεν έπρεπε να έχει γίνει η επέμβαση στη Λιβύη, αλλά λέω ότι στο επίπεδο της ε, επέμβασης στη Λιβύη προσπαθήσαμε να ε, κάνουμε την απαιτούμενη συγκράτηση της κατάστασης. Εκατοντάδες αντάρτες πήγαν στη... στο Μαλί και αλλού βέβαια. Και εγώ τότε είχα μιλήσει με φίλους που ήταν κοντά σε αυτή τη διαδικασία λήψη αποφάσεων και μα έλεγαν δεν έχουμε εξουσία για να παρέμβουμε στα σύνορα. Αυτό τι θα πει, ότι παρόλα αυτά σε αυτή την περιοχή του κόσμου και πραγματικά το, το Μαλί είναι εμβληματικό. Έχουμε μια μετατόπιση κινδύνων παντού. Θα το δούμε με τρομοκράτες ε, που πάνε ε, προς την Αλγερία, Μπουρκίνα Φάσο κτλ. Είναι πάρα πολύ ε, ρευστά τα πράγματα σε αυτή την περιοχή στρατηγική για το Σαχέλ ε, ήταν μια επιτυχία της Ένωσης, το 2011 την καταρτήσαμε, αλλά έχουμε ασχοληθεί περιφερειακή ανάπτυξη, καταπολέμηση λαθρεπών υποτικών Σαχέλ, στο Σαχέλ. Κάπως τα είχαμε δηλαδή προβλέψει όλα αυτά, αλλά αυτή την ιδέα της μετατόπισης του κινδύνου σήμερα είναι δύσκολο κανείς να ε, προβλέψει τι μπορεί να γίνει και μετά θα έχουμε εξάπλωση από το μαλλί αλλού. Εγώ πιστεύω ότι πρόκειται ουσιαστικά για νέους πολέμους που ζούμε. Νέα είδος επίθεσης. Νέα είδη επιθέσεων πρέπει να κάνουν. Αυτό που είπες για τις εκλογές είναι μια ιδέα που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Αλλά νομίζω ότι βλέπουμε μόνο το, την κορυφή του παγόβουνου. Αυτό έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής μόνο. Επειδή όμω υπάρχει ζήτηση για ναρκωτικά, ε, για εμπορία ανθρώπων, θα δούμε να μετατοπίζονται, να μεταφέρονται οι τρομοκρατικές ομάδες και εκεί δεν έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο και αυτό με ανησυχεί. Καθένας έχει τις δικές του ε, εντυπώσει. και τώρα διαφορώ πλήρω αν ο Σαρκοζή έπαιξε το χαρτί τη Λιβύη και άρα ο Λάντε πρέπει να παίξει το χαρτί του Μαλί και ούτω καθεξή. Εδώ και ένα χρόνο ζητούσαν βοήθεια και μετά κινήθηκε η Γαλλία. Αυτό το είδαμε, το είμαστε μάρτυρες. Τώρα, το δεύτερο, Αφιλέσω στο ερώτημα, εγώ συμφωνώ μαζί σου για αυτόν τον α, στρατιωτικό. Αυτός είναι νέος, σχεδόν έγινε αρχηγός κράτους και δεν θα τα καταλήψει εύκολα, θα τα παρατήσει. Τι θα κάνει και εν ώψη μελλοντικών εκλογών τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει να μην παίξει ο Σανόκο. Ποια σχέση θα μπορούσε να έχει με τις εκλογές, πώς θα ήταν ανησυχητική η ενδεχόμενη μπλοκή του. Νέα είδη πολέμου λοιπόν, δεν έχουμε λάμψει μέχρι τώρα και το ειδικό πρόβλημα, τα ειδικά προβλήματα, ειδικά για το μαλλί εννοώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκέρνς τώρα έχει το λόγο. Δεν θα ήθελα να, πάρα, να είμαι πολύ αυστηρός με τη Γαλλία. Η Βερονίκ το επενθύμησε. Είχε ζητήσει βοήθεια το Μαλί και μόνο όταν έγινε προφανές ότι η φόρμουλα που είχε βρεθεί στο επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας δεν λειτουργεί, γιατί οι ενοπλές δυνάμεις των κρατών μελών της οικονομικής κοινότητας της ε, Δυτικής Ευρώπης δεν ήταν έτοιμες, τότε μόνο επενέβη η, επενεύει Γαλλία, γιατί δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική. Μπορούμε να διερωτηθούμε για το τι ε, υπήρχε στο μυαλό των μεν και το δε από πίσω. Γιατί κάποιοι εγωισμοί υπάρχουν, εντάξει, αλλά οι αλτουριστές υπάρχουν και αν υπάρχουν που είναι. Οι πιο πολλοί ήταν οι αδιάφοροι τελικά. Έτσι ήταν η κατάσταση. Ξέρουμε ότι δεν είναι τέλεια τα πράγματα. Αυτό που με ανησυχεί εμένα είναι ότι τελικά δύσκολα μπορεί κανείς να διακρίνει μια βιώσιμη λύση. Στην περιοχή του Κιντάλ που τη γνωρίζω, είδαμε τι έγινε. Νομίζω ότι μόνο αν υπάρξει ανάληψη ευθύνης των του ΑΡΕΓ, αν ε, ε, αναλάβουν τις ευθύνες που είναι και το δομικό στοιχείο της περιοχής του ΑΡΕΚ, θα έχουμε μία βιώσιμη λύση. Σε κάθε επίπεδο πρέπει να αναλυφθεί ευθύνη και στο επίπεδο της κυβέρνησης, ε, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, είναι μία δυνατότητα που πρέπει να εξεταστεί και ε, έχει δίκιο ο Λουί Μισελ, τον οποίο και συγχαίρω για την εξαιρετικά διευγή ανάλυση του, ότι πράγματι πρέπει να έχουμε περιφερειακές λύσεις. Ανέφερε επίσης τα πραγματικά προβλήματα που θα προκύψουν η Βερονίκη Ζερ και νομίζω ότι η απάντηση είναι ακριβώς η πρόθεση περιφερειακής διάστασης. Οι Αφρικανοί εμπνέονται από το ευρωπαϊκό μοντέλο που δεν λειτουργεί όμως και αυτό είναι πραγματικά κάτι που μας ε, συγκινεί. Δεν λειτουργεί όμως το ευρωπαϊκό μοντέλο. Οι ελπίδες μας βασίζονται σε αυτούς που είναι έτοιμοι να λάβουν τις ευθύνες τους. Εκεί που η Ευρώπη όμως είναι ανίκανη να δράσει. Άρα τώρα τιμάμε το εξή. Δεν ξέρω αν εσύ τη δυνατότητα, Λουί, να δώσεις κάποια απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα στο Μαλί. Χρονικά, πότε πιστεύω ότι θα μπορούσε θα μπορούσαν οι ένοπλε δυνάμει περιοχή να αναλάβουν ευθύνε. Ξέρουμε ότι είναι το τσάντ παρόν, ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα ανεφοδιασμού. Ποιο ασχολείται, ποιο προσπαθεί να επιλύσει αυτά τα προβλήματα. Αυτό νομίζω θα ήταν δυνατό να τα προβλήματα αυτά τα λύσουν οι ίδιοι Αφρικανοί με την ε, βοήθεια, τη διοικητική μέρη από πλευρά Ένωση. Αυτό θα ήταν η αρχή όμως. πρέπει να υπάρξει αυτή η διάρθρωση μιας πολιτικής επιχειρησιακής απάντησης στην περιοχή. Και αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί με μια πάρα πολύ ισχυρή εταιρική σχέση της περιοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο τώρα στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στον κύριο Πιέρ Κριστόφ Χατζησάβα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Προέδρε. Αν επιτρέπετε, θα ήθελα να επιθυμίσω εν ολίγη τις αποφάσεις που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση συλλογικά και μεμονωμένα τις τελευταίες εβδομάδες και μετά θα αναπτύξω και κάποια σημεία που ήδη εφήγησαν στη συζήτηση συμπεριλαμβανομένης περιφερειακής διαστάσεως και της στρατηγικής για το Σαχέλ. Από τα ανάρχησαν δικές επιχειρήσεις 10 και 11 Ιανουαρίου Πιο συγκεκριμένα μετά την έγκριση οδικού χάρτη μεταβατικού τέλος Ιανουαρίου από την κυβέρνηση του Μαλή και την Εθνοσυνέλευση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε κάποιες αποφάσεις που συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε και θα επιταχύνουμε την εφαρμογή του Εν πρώτης, στον τομέα της ανάπτυξης, τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να επαναληφθεί σταδιακά η αναπτυξιακή βοήθεια, οπότε βραχυπρόθεσμα θα εγκριθεί ένα πακέτο δράσης ύψους περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ, δημοσιονομική υποστήριξη πάρα πολύ σημαντική. Ε, στόχος είναι να βοηθήσουμε την κυβέρνηση του Μάλι να αποκαταστήσει την εξουσία του όλη την επικράτεια, την εξουσία της όλη την επικράτεια και να αποκαταστήσουμε τη δυνατότητα της κυβερνήσης να παρέχει δημόσιες υπηρεσίες βασικές στις περιοχές που απελευθερώθηκαν από την τρομοκρατική κατοχή. Παράνοιμα, υιοθετήσαμε διάφορα μέτρα όσον αφορά το μέσο σταθερότητα, σταθεροποίηση μάλλον, για να εφαρμοστούν δράσει σε διάφορου τομεί, όχι πρόθεσμα. Συμπεριλαμβάνεται η σταθεροποίηση, η προετοιμασία εκλογών, ε, ενίσχυση για τι δυνάμει ασφαλεία, δηλαδή για την διατήρηση τη τάξη και την καταπολέμηση τη εγκληματικότητα. Αυτά για την αναπτυξιακή πτυχή. Όσον αφορά την ασφάλεια, για αυτή την πτυχή, Κάποιοι ομιλητέ ήδη αναφέρθηκαν στην υποστήριξή μα στην αποστολή την Αφρικανική για την σταθεροποίηση στο Μαλί. πρόθεσμα είναι η προσέγγιση. 50 εκατομμύρια ευρώ ε, δεσμεύτηκε να δώσει ο Επίτροπο ε, Πίμπαλ στι 29 Ιανουαρίου σε μια συνεδρίαση ε, των δωρητών. Μετά έχουμε τις πληρωμές αποζημιώσεων στους στατιώτες που είναι επιτόπου και τους στρατιώτες του Τσάντ που είναι υπό την ε, ηγεσία ε, της Αφρικανικής Ενώσεως. Αυτά τα χρήματα, τα 150 εκατομμύρια θα δοθούν στο στρατό του Μίσμα μέσα Απριλίου το αργότερο, αλλά η χρηματοδότηση είναι αναδρομική. Και αυτό το μήνυμα το επιβάσαμε σε όλες τις χώρες ε, που συμβάλλουν με στατεύματα υπό τις περιστάσεις που ενθυμίστηκαν. Δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν προβλήματα επιχειρησιακά, επιμελητιακά, τα αφρικανικά στρατεύματα είναι 6.200 αριθμό, 2.000 από αυτούς είναι από το Τσάντ. Σημαντικός αριθμός στρατευμάτων, ε, παίζουν ρόλο σημαντικό οι στρατιώτες και θέλουμε να αυξηθούν τα στρατεύματα τις επόμενες εβδομάδες να φτάσουμε στους 9.500 στρατιώτε. Άρα η υποστήριξη της Ευρωπαϊκή Ενώσεω δεν είναι μια υποστήριξη η οποία είναι προβλέψιμη και που επαρκεί όσον αφορά τη διάρκεια. Άρα Κατεπηγόντω πρέπει να θετηθεί ένα ψήφισμα από το Συμβούλιο Ασφαλεία, ώστε να μεταμορφωθεί αυτή η αποστολή σταθεροποίηση σε αποστολή ε, σταθεροποίηση και εξασφάλιση τη ασφαλεία από πλευρά του ΟΗΕ. πρόθεσμα επίση και στον τομέα τη ε, ασφάλεια η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε μια αποστολή η οποία δεν θα μπορούσε να δει το φως της ημέρας χωρίς δέσμευση από πλευράς κρατών μελών, μεμονωμένα και συλλογικά η αποστολή θα μπορέσει να ασχοληθεί με την εκπαίδευση των στρατιωτών του Μαλή εντός των προβλεπωμένων προθεσμιών, διότι τα κράτη-μέλη στο σύνολό τους σε αυτή την αποστολή έστειλαν τα στατεύματα που απαιτούντο και τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν την επιχείρηση αυτή την ευρωπαϊκή. Είναι σημαντικό να αναφερθεί. Τέλος, όσον αφορά τον πολιτικό τομέα, υιοθετήθηκε ο δικός χάρτης υιοθετήθηκαν κείμενα που θα ρυθμίζουν την θέσπιση αυτή τη Επιτροπή Εθνική για τη συμφιλίωση και το διάλογο και από αυτή τη βάση αποφασίσαμε ξαναρχίσουμε τον πολιτικό διάλογο με την κυβέρνηση 18 Φεβρουαρίου και αυτό δείχνει εμβληματικά τη θέση μα. Αναγνωρίζουμε τη μεταβατική κυβέρνηση σαν την νόμιμη αρχή του Μάλι. Θεωρούμε ότι αυτή η κυβέρνηση και ο πρόεδρο ο πρόεδρο Τραωρέ αντιπροσωπεύει τη συνταγματική συνέχεια και θεωρούμε ότι μπορούμε να ξαναρχίσουμε τον πολιτικό μας διάλογο χωρίς να προσφύγουμε όπως τον περασμένο χρόνο στο άθρο 96. Κάποιες λεπτομέρειες στον αφορά τις επιχειρησιακές στοιχές οι οποίες αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των προτέρων ανταλλαγών απόψεων. Λοιπόν, οι βιοπραγίες από πλευράς του στρατού του Μάλι Όλοι είμαστε πολύ ευαίσθητοι όσον αφορά αυτές οι εικασίες για αυτές τις πράξεις που έλαβαν χώρα σε απελευθερωμένες περιοχές του Μάλι. Είναι μια πτυχή είναι κασίες ή πραγματικά περιστατικά που υπονομεύουν το διάλογο και σταθερότητα του Μάλι μακροπρόθεσμα και γι' αυτό γίνονται διαβουλεύσεις και μεμονωμένα κάποια κράτη μέλη που είναι παρόντα στο Μάλι επισκέπτονται εκεί κάνουν συνομιλίε με τι τόπιε αρχέ, αλλά και συλλογικά η Ευρωπαϊκή Ένωση το ζητά αυτά δυνάμει του άρθρου 8 του, άρθρου, του Κοτονού, τη Συμφωνία Κοτονού que euh, la επιμείναμε η διεθνής κοινότητα να αναπτύξει το ταχύτερο δυνατόν εκεί παρατηρητέ. Η Αφρικανική Ένωση δεσμεύτηκε να το κάνει με την υποστήριξή μα. Επίση, θέλουμε και ανεξαρτήτου παρατηρητέ τη κοινωνία των πολιτών, κάτι που θα γίνει τι επόμενε εβδομάδε. Όσον αφορά τι εκλογέ. Το χρονοδιάγραμμα για τι εκλογέ πραγματικά είναι γνωστό. Είναι προστατευμένο στον οδικό χάρτη στον οδικό χάρτη που υθετήθηκε από την κυβέρνηση και την συνέλευση του Μάλι. Στόχο είναι να διεξαχθούν εκλογέ το μήνα Ιούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται, δεσμεύτηκε και θα δεσμευτεί να δώσει εκλογική αρρωγή για να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Επίσης θα αποστείλουμε εν ευθέτω χρόνο μια αποστολή διερευνητική για να, ε, στείλουμε εκεί και παρατηρητέ για την εξαγωγή των εκλογών. Είναι σαφέ και το επεθύμησα κατά κάτι μέλη στο προηγούμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ότι ο σεβασμό του χρονοδιαγράμματο που καθορίστηκε από τον οδικό χάρτη είναι ένα στοιχείο θεμελιώδε για την αξιοπιστία τη διαδικασία τη μεταβατική στο σύνολό τη. Λοιπόν, θεωρούμε για την ώρα ότι ο σεβασμό και η τήρηση του χρονοδιαγράμματο, πιο συγκεκριμένα του στόχου τη διεξαγωγή των εκλογών το μήνα Ιούλιο, είναι σημασία για τη σταθερότητα και για τη διαδικασία τη μετάβαση εν γέννη. Τέλος, όσον αφορά το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο υπογραμματέας ο κ. Μιούλιτον του ΟΗΕ, πήγε στο Μαλί σε αποστολή την περασμένη εβδομάδα. Θα παρουσιάσει με έκθεση το Συμβούλιο Ασφαλείας στις 25 Μαρτίου. Και οι διαβουλεύσεις που θα απορρεύσουν από αυτή την παρουσίαση θα επιτρέψουν την οθέτηση ενός ψηφίσματος που θα δημιουργεί μια αποστολή σταθεροποίηση μέχρι μέσα Απριλίου. Και τέλος, Όσον αφορά τα, την περιφερειακή πτυχή, υπενθυμίσαμε εδώ την ύπαρξη στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το Σαχέλ, για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στο Σαχέλ. Αυτό το μέσο ήταν θεμελιώδου σημασία για να δημιουργηθεί συνένεση ευρωπαϊκή, να υπάρξει αντίληψη ευρωπαϊκή για το τι γίνεται με την κρίση αυτή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να κινητοποιηθούν συμπληρωματικοί πόροι μέσω του ΦΕΔ αλλά και μέσω του μέσου σταθεροποίηση θα υποβάλουμε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων μηνό Απριλίου μια έκθεση για την εφαρμογή των λόγων στρατηγικών, αλλά ήδη είναι σαφές ότι τα κράτη-μέλη μας, όπως μας εκάλεσαν στο προηγούμενο Συμβούλιο, μας κάλεσαν να η εφαρμογή και υλοποίηση στρατηγικής και σε το εγκύτατο μέλλον θα δούμε πώ μπορούν να επεκταθούν οι δραστηριότητε στρατηγική σε διάφορε χώρε, οι οποίες εξίσου επηρεάζονται από την περιφερειακή κρίση συμπεριλαμβανομένου του Μπουρκίνα Φάσου, του Τσάντ και τη Σενεγάλης. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Λουί Μισελ, έχετε το λόγο για να κλείσετε. Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Ε, ξέρετε, δεν θέλω να εμβαθύνω ε, όσον αφορά την ψυχολογία που οδήγησε στην παρέμβαση της Γαλλίας Λυπούμε, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό. Συστηματικά όταν μια χώρα πάει στην Αφρική, ευρωπαϊκή χώρα πάει στην Αφρική, εδώ είναι η Γαλλία, αμέσως υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει τα στα κίνητρα και τα έτια αυτή η χώρα. Γιατί εγώ είμαι αρκετά αφελής, κυρία μου. Έχω την αγνότητα του αφελούς. Νομίζω ότι τα κίνητρα του κυρίου Ολάντ είναι αγνά κίνητρα για να το πω μα και δεν με νοιάζει κασίλα μου. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ξέρω κατά πόσο αυτή η συνεισφορά, αυτή η πρωτοβουλία της Γαλλίας θα αλλάξει τα δεδομένα. Και αυτό κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί. Ότι αλλάζει ριζικά τα δεδομένα. Εάν υπήρξε κάποια συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αυτής καθεαυτής σε αυτή την περιοχή θα μπορούσαμε να σπάσουμε τη ραχοκοκαλιά του φονταμεταλισμού του επικινδύνου φονταμεντελισμού που πάει να αναπτυχθεί σε όλη αυτή την περιοχή. Και θα ρυθμίζει και το πρόβλημα αυτό τη ε, μετακίνηση του προβλήματο που αναφέρατε, διότι περί αυτού πρόκειται προφανώ. Εγώ θέλω να πω ότι όσον αφορά. Α, το άλλο. Α, να πω κάτι, κάτι του Αρέγ. Ξέρω ότι χαλιναγωγήθηκε το θέμα των του Αρέγ, το καταλαβαίνω, είναι κάτι. Ε, είναι μια μειονότητα, κάθε μειονότητα δημιουργεί συναισθηματισμό των γενναιοδόρων. Όλοι είμαστε γενναιόδοροι άνθρωποι με καλές προθέσεις. Η τουαρέγκ είναι κάτι, κάτω το 2% του πληθυσμού του Μαλή. Να το επιθυμίσουμε. Το πρόβλημα των Τουαρέγ οι Τουαρέγ έχουν στο Κιντάλ έχουν 85% πλειοψηφία. Αλλού είναι στη μειοψηφία, αλλά έχει στη μειοψηφία. Και στο Κιντάλ υπάρχει ένα πρόβλημα. Πολιτισμικό-ιστορικό πρόβλημα η κοινωνία των Τουαρέγ, ας πούμε, πώς να το πούμε, το κόρπους, ο κορμός του Αρέγ εδράζεται επί θεοδαλικής ιεράρχησης. Δεν, μην το παίρνετε έστραβα αυτό, εγώ δεν θέλω να προσβάλλω, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Φιλετικό και σε κάστες βασίζεται. Περιπλοκότατο. Τι να σας πω το δεν το καταλαβαίνετε στο Κιντάλ. Ακούστηκαν καταγγελίε κατά τη Γαλλία για το Κιντάλ. Οι Γάλλοι προσπαθούσαν να πάρουν το Κιντάλ ήπια, προσπαθώντα να έρθουν σε διαλόγο με το MLA, που είναι δημόσιο κίνδυνο υπαριθμών 1. Για το MNLA ε, είναι γύρω από το Κιντάλ μία οικογένεια του ΑΡΕΓ που έχει την εξουσία στο Κιντάλ και θέλουν να διατηρήσουν την εξουσία και τσακώνται με άλλη οικογένεια που θέλει να την καταστήσει Πολύ περίπλοκα, πολύ περίπλακα τα ζητήματα του ΑΡΕΚ. Δεν νομίζω. Τι να σα πω. Τέλο όσον αφορά τι δράσει κατά τον του ΑΡΕΚ, δεν θα επανέλθω. Πρέπει να σας πω ότι αν θέλετε ο Σανάκο να ξαναπάρει το, την εξουσία στο Μάλι θα πρέπει να κάνουμε αυτό που προτείνατε, να καθυστερήσουν, να δημιουργηθεί μια συντακτική συνέλευση μια συνταγματική συνέλευση πώς θα είναι πιο ηθική από εκλογές. Δεν καταλαβαίνω. Θα απαρτίζεται η συνέλευση από εκπροσώπους που θα έχουν καθοριστεί χωρίς καμία νομιμότητα. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλύτερα να διοργανωθούν το ταχύτερο δυνατόν εκλογές. Είχα κάποιες αμφιβολίες αφορά τη δυνατότητα διοργάνωση εκλογών στη συνεδρίαση με το Διευθυντή των Εκλογικών Υποθέσεων, με τον Υπουργό της Περιφερειακής Διοίκησης, Εδαφικής Διοίκησης και του άλλους αρμοδίους, ε, με καθησύχασαν. Διότι ε, έχει γίνει η καταγραφή, ε, οι εκλογέ έχουν καταχωρηθεί, υπάρχει καταχώρηση βιομετρική, καλά έγινε, το μόνο πρόβλημα παραμένει πώς θα διοργανώσουν την ψηφοφορία από πλευράς των προσφύγων και των εκτοπιστέντων. Αν γίνουν προεδρικέ εκλογέ, εντάξει. Αν γίνουν αμέσω οι κοινοβουλευτικέ εκλογέ, υπάρχει πρόβλημα. Το πρώτο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα. Πολλές... Δεν υπάρχει τοπική αυτοδίκηση παντού. Προσπαθούν να αποκατασταθεί α, και χρειάζεται αυτή η προσπάθεια. Ρωτήσατε μήπως και σωστά το Μάλι εθεωρεί το καλό παράδειγμα στην Αφρική. Ομόφωνα. Εγώ δεν το είχα δει έτσι. Λέμε σήμερα ότι ήταν μια δημοκρατία εικονική, πρόσωψη δημοκρατίας. Τυπικά, με εναλλαγές κλπ. Να πω κάτι και μετράω τα λόγια μου. να δούμε πώς θα συμπεριφερθούν άλλε χώρες, όπως η Αλγερία και η Μαυριτανία, που σε όλα αυτά τα ζητήματα έχουν περίεργη στάση. Δηλαδή συγκράτηση ένοχή θα έλεγα. Τώρα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Δύσκολο να έχουν αόριστη στάση. Αντικειμενικά που το βλέπω από πολύ καιρό, θεωρώ ότι αυτό χρειάζεται εμβάθυνση. Ειλικρινά, αν υπάρχει προτεραιότητα για μένα, χρειάζονται εκλογές ταχύτερο δυνατόν. Αυτή είναι η προτεραιότητά μου. Και δεν θα γίνουν 100% τέλειες εκλογές. 90% θα είναι τέλειες ίσως. Αυτό που είναι σημαντικό είναι οι πρόσφυγες και εκτοπιστέντες να συμμετάσχουν. Διότι αν περιμένουμε θα δοθεί χρόνος σε όλες τις αρνητικές δυνάμεις να κινηθούν. Άρα θα πέσει εν κενό, σε κενό η γαλλική πρωτοβουλία να το κάνουμε αυτό. Μετακίνηση του κινδύνου, συμφωνώ βέβαια. Βερονίκ, το θέμα αυτό το ξέραμε. Στην ε, ισομερή συνέλευση δεν το συζητούσαμε το πρόβλημα αυτό και ξαφνικά μας δεν θα δείτε ότι θα έχουμε πρόβλημα. Διότι γνώριζαν τότε ότι ήδη υπήρχαν ε, κάποιες ε, συμμαχίες μεταξύ των λαθρεμπόρων ναρκωτικών, των εμπόρων ε, λευκής αρκός, των ανθρώπων, των φοντεμετελιστών και ήξεραν ότι το πρόβλημα έρχεται. Στατική για το Σαχέλ. Δεν θα ρυθμίσουμε τίποτα αν δεν εφαρμόσουμε μια γενική στατική για όλη την περιφέρεια αυτή το είπα. Όσον αφορά... Α, ο Σάλμας θέτει ένα ερώτημα. Πότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι ο στρατός του Μάλι θα μεταρρυθμιστεί παρκώς για να μπορεί να λειτουργήσει. Είναι σημαντική οργάνωση. Η ΣΕΝΤΕΑΟ, λοιπόν, τι να σας πω, δεν σας μήνυσα. Σκόπιμα γι' αυτό, αλλά μου το θέσατε. Η ΣΕΔΕΑΟ, τι να πω, είναι κάτι πολύ σημαντικό, σημαντικό για να την υποστηρίξουμε, να την αξιοποιήσουμε, αλλά κινείται σαν να μην ήταν η Γαλλία που κάνει τη διαφορά. Ότι θα κάνει τα πάντα, αυτό διαφημίζεται. Αλλά πώς, χρειάζεται μέσα θα ήθελε να αντικαταστήσει μια διεθνή κοινότητα που είναι λιματική. Μόνη τη Γαλλία δεν μπορεί να κινηθεί. Μπορεί να τα καταφέρει, χρειάζεται εξοπλισμός, πρέπει να χρηματοδοτηθεί αυτό που εν μέρει γίνεται και χρειάζεται και κατάρτιση. Θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο. Χρειάζεται χρόνος για να εκπαιδευτεί ο στρατός του Μάλι είπαν ότι ο στρατό δεν έκανε αυτό που έπρεπε. Δεν είναι γιατί δεν έγινε σωστή μετάχυση του στρατού. Όπω λέω εγώ τα πράγματα. Για να επιτεθούμε κατά των αιτίων, όπως το θέμα των του ΑΡΕΚ δεν πρέπει να μιλάμε για φεντεραλισμό, όμως μπορούμε να μιλάμε για αποκέντρωση με χρήσιμο τρόπο, διότι η αποκέντρωση ναι θα είναι μια λύση. Όλη η περιοχή του Κιντάλε θα μπορούσε να αναπτυχθεί, κυρίως στον τομέα της γεωργίας. Έχουν πρόβλημα, όλη αυτή η περιοχή του βορρά θα πρέπει να απεγκλωβιστεί. Θα πρέπει η ανάπτυξη να βασιστεί στην επικοινωνία, στην συγκοινωνία και εντός της χώρας, εντός Μάλι και σε επικοινωνία και με τη χώρα. Προσπάθησα να απαντήσω κυρία Πρόεδρε. Μπορούσα να μιλήσω πολύ Θα δώσω την άδεια στην κυρία Γκρέσ να κάνει μια σύντομη παρέμβαση. Κυρία Γκρέσ, ναι, μάλλον δεν με κατανόησε πολύ καλά ο κύριο Μισελ. Εγώ δεν είπα ότι η κατάσταση θα ήταν καλύτερη αν δεν είχε επέμβει η Γαλλία. Δεν είπα αυτό. Ε? Θα ήταν χειρότερη από ό,τι είναι σήμερα στον Παμάκο. Αυτό που είπα και το επαναλαμβάνω γιατί απάντηση δεν πήρα σε αυτή τη συζήτηση, είναι ότι στρατιωτική λύση συνεκλογές δεν θα λύσει το ζήτημα της ανάπτυξης και της στόχιας στο Μαλί, γιατί αυτό οδήγησε σε αυτή την κατάσταση, αυτό το πρόβλημα. Νομίζω δηλαδή ότι τα ίδια αίτια θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε ε, στην ε, κάθαρση, αν θέλετε, ε, των ε, πληθυσμών και να νομίζουμε ότι ξεκινάμε από το μηδέν. Αυτό ήθελα να πω. Αν ε, κάποιο έχει πυρετό μπορούμε να σπάσουμε το θερμόμετρο, αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Λουί Μισελ. Μα τι να σας απαντήσω, ε, σε ρητορικά ερωτήματα τι να απαντήσω. Φυσικά και έχετε δίκιο, σας, ε, δίκιο κυρία μου, δεν είπα εγώ ότι οι εκλογές ή ε, αν εκαθαρίσουμε ε, τους φονταμεταλιστές αυτό θα την καταστήσει την ανάπτυξη, είναι όμως προεπαιτούμενο. Αν δεν υπάρχει μια πολιτική σταθερότητα στοιχειώδης, και ε, ασφάλεια στοιχειώδης, τι ανάπτυξη να υπάρξει. Είναι απλά τα πράγματα, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Εγώ, ακούστε, θα απαντήσω ε, με κάτι παράλογο αν θέλετε. Να φανταστούμε σήμερα το Μαλί ή όλη την ευρύτερη περιοχή. Πώς θα ήταν σήμερα, εάν δεν είχε επέμβει η Γαλλία, Νομίζω η απάντηση στο ερώτημα αυτό απαντάει και στο δικό σας ερώτημα. Για το εκαθάριστο φανταμεταλιστών, ναι εντάξει, ξέρετε όμως πρέπει να πάει κανεί και επιτόπου για να δει τι γίνεται. Όταν αυτοί επιβάλλουν ε, τη σαρία που κόβουν χέρια, αν δείτε πώς φέρονται στις γυναίκες, ε, είναι απίστευτη συμπεριφορά. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν. Πάντως μαζί σας συμφωνώ και γι' αυτό συζητήσαμε για την ανάπτυξη. Δεν είχα το λόγο χρόνο να το θέσω εγώ το θέμα αυτό της ανάπτυξης, αλλά έχουμε τα ζητήματα υποδομών, μεταφοράς τεχνολογίας στη γεωργία κτλ. Όλα αυτά τα είπαμε. Φυσικά συμφωνώ ότι χρειάζεται ένα σχέδιο και σε αυτά τα θέματα. Πρόεδρος, θα μπορούσαμε να μιλάμε επί ώρες ακόμα για το Μαλί. Άφησα να ξεπεράσουμε πάρα πάρα πολύ το χρόνο μας αφού ε, για μια φορά είχαμε μια πάρα πολύ συναρπαστική, σημαντική συζήτηση για μια φορά ή για ακόμα μια φορά. Και ξέρετε, χαίρομαι και που έχουμε τόσους συμμετέχοντες, γιατί ήταν λίγοι πολλές φορές συμμετέχοντες. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για το Μαλί. Ο κύριος Μπέρμαν μου έχει ζητήσει το λόγο για δύο-τρία λεπτά. Γιατί έχει μία ανακοίνωση να μας κάνει ο κύριος Μπέρμαν για το DCI οχι δύο 2-3 λεπτά, 30 δευτερόλεπτα, λέει ο κύριο Μπέρμαν. Παίρνετε συνδρές και κλεισμένο των θήρων για τον DCI. Όχι. Α, λέω κι εγώ. Λοιπόν, 30 δευτερόλεπτα να σας πω ότι εμείς στο Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσει για το DCI, δηλαδή για το μέσο μεταξύ συνεργασίας, δεν θέλουμε χρόνο, γιατί είναι σαφή τα αιτήματά μας ε, και το τι επιθυμούμε είναι πολύ ξεκάθαρο. Το Συμβούλιο είναι αυτό που μας κάνει να χάσουμε χρόνο. Με αυτή την έλλειψη σαφήνεια που δύσκολα μπορούμε την αποδεχτούμε, πρέπει να διαπραγματευτούμε, πρέπει να βρούμε λύση και διέξοδο για να προγραμματίσουμε, γιατί πρέπει μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2013 να συνεχιστεί η αναπτυξιακή βοήθεια. Η Κομισιόν πήρε το χρόνο που ανάγκη για να φτιάξει αυτό το πολύ χρήσιμο non-paper, ήρθε μεν με καθυστέρηση αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο, είναι η βάση για τι τι περιμένει το Συμβούλιο. Avec nous. Tout ce que je veux dire. Merci. Τι περιμένει το Συμβούλιο για να προχωρήσει μαζί μας. Αυτό είχα να πω. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ και εισηγητά, για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε στο σημείο 17 της ημερησίας διάταξης. Contre la fraude fiscale που είναι η καταπολέμηση της ε, φοροαπάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων. Δαπανίσαμε πολύ χρόνο ήδη. Λοιπόν, ας δώσουμε και πέντε λεπτά για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Να μιλήσω πρώτα εγώ, αφού είμαι και η συγγήτρια. Η συγγήτρια ουσιαστικά συντάγρα της γνωμοδότησης. Θα ξέρετε, ορισμένοι από εσάς, πόσο με ενδιαφέρει και εδώ και πόσο καιρό με ενδιαφέρει αυτό το θέμα και δεν είναι τυχαίο, το είδαμε και σήμερα το πρωί. Είδαμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα. Είναι εξίσου σημαντικό τα τελευταία χρόνια, ίσως και περισσότερο. Ένα, δισεκατομμύριο, ένα τρισεκατομμύριο περίπου είναι οι απώλειες ετησίως που έχουν τα κράτη-μέλη λόγω της φοροδιαφυγής 2.000 ευρώ ανά Ευρωπαίο πολίτη. Και για μας αλλά και για τις στοχές χώρες αυτό συνιστά ε, τροχοπέδι στην ανάπτυξη. Επίσης, υπάρχει το πρόβλημα των ε, παράνομων ε, χρηματοοικονομικών ροών. Σήμερα το πρωί είχαμε τον Raymond Baker από την Global Financial Integrity που μας υπενθύμησε ότι μιλάμε για περίπου 8 δολάρια παράνομων ροών για ένα δολάριο που εμείς στέλνουμε και εκπονεί αυτή η οργάνωση μια νέα μελέτη τεκμηριωμένη, πληρέστατη και τα αποτελέσματά της δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν μειώνεται. Τι σημαίνουν αυτά όλα σημαίνουν ότι οι φτωχές χώρες συνεισφέρουν 10 φορές περισσότερο στην οικονομία των αναπτυγμένων χωρών από ότι ε, η βοήθεια που τους δίνουμε εμείς. Επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Γαλλία και η Νορβηγία σήμερα χρηματοδοτούν μια μελέτη του ΟΣΑ για τη δημιουργία μιας ειδική ε, ε, ομάδας δράσης ε, Task Force για την παροχή βοήθειας στις χώρες αμψόμενες ώστε να μπορέσουν να εντοπίσουν τη φοροδιαφυγή και να έχουν και περισσότερους ίδιους πόρους στη διάθεση τους. Στόχος επίσης είναι η ισότιμη και πιο δίκαιη φορολόγηση. Η ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών είναι ένας παλιός αγώνας που δίνουμε στην οδηγία περί αποταμιεύσεων Savings Directive. Έχουμε συμπεριλάβει αυτή τη ρήτρα για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πρέπει να υπάρχει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των χωρών. Και αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε στο πλαίσιο μιας πολυμερούς δεσμευτικής συμφωνίας. Χαιρετίζω τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέλει να προχωρήσει με αυτή την αυτό με την ανταλλαγή πληροφορίων. Ο δρόμος που έχει επιλέξει ο ΣΑΤ, ο διμερής δηλαδή, αυτός δρόμος ουσιαστικά είναι μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης. Είναι λόγος της ύπαρξης αυτών των συμφωνιών. κάνουν forum shopping οι εταιρείε, διαλέγουν τις συνθήκες ε, για να μπορέσουν να βελτιστοποιήσουν τα κέρδη τους και βέβαια βελτιστοποιούνται και μεγιστοποιείται και η φοροαπάτη και φοροδιαφυγή σε παγκόσμια κλίμακα. Θα έχουμε το country by country reporting, αναφορές εκθέσεων αναχώρα, για να έχουμε περισσότερη διαφάνεια. Και σήμερα το πρωί ακούσαμε για το εμπορικό σκέλος ε, των παράνομων οικονομικών ροών. 65% των ροών για το 65% είναι υπεύθυνες πολυεθνικές. Έχουμε διαφθορά 5% και 30% τόσο είναι το έγκλημα ευρύτερα. Κλιματικές δραστηριότητες. Θα πρέπει επίσης να θεσπίσουμε μητρώα για τα ιδρύματα και για τα τράστε Θα, θα πρέπει να δούμε να ξέρουμε με ποιους συναλλασσόμαστε. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπάρχουν διατάξεις που θα είναι το αντίστοιχο, το ισοδύναμο της ε, πράξης Dot Frank στις ΕΠΑ. Δηλαδή, θα απαγορεύσουμε τις εταιρείες ε, που δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιοι, είναι, τα, τα, ποιοι είναι τα τελικά φυσικά πρόσωπα δικαιούχοι. έχω περιορισμό θα κάνω και τροπολογίες για να συμπληρώσουμε την, ε, την έκθεση. Ξέρετε ότι έχουμε κάποιο περιορισμό με, τα, με τις γραμμές, ε, με το πόσους χαρακτήρες μπορεί να έχει μια γνωμοδότηση. θα δούμε, θα το διορθώσουμε αυτό. Αυτά είναι τα πλέον ε, προεξάρχοντα ζητήματα για το θέμα αυτό η Κομισιόν δεν ε, διαφωνεί. Άρθρο 50. Λοιπόν, δεν βλέπω να θέλει κανείς να λάβει το λόγο. Είναι ένα θέμα για το οποίο συζητήσαμε διαμακρόν άλλωστε και σήμερα το πρωί. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mm. Τρεις βλέπω ότι είστε εκεί. Διαλέξτε. Διαλέξτε ποιος θέλει να λάβει το λόγο. Αλλιώ θα θεωρήσω ότι συμφωνείτε απόλυτα μαζί μου. Και ότι η νομοθεσία που περιμένουμε το φθινόπωρο θα περιλαμβάνει αυτά τα στοιχεία, δηλαδή την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, αυτόματο mm. μητρό, country by country report. Έχετε το λόγο. Thank you very much, Madam President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίσουμε βεβαίως ε, την ε, ε, τον ενδιαφέρον που δείχνει η Επιτροπή Ανάπτυξης για την πρόταση της Κομισιόν, για την φοροαπάτη και τη φοροδιαφυγή και την αντιμετώπιση τους. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν περιορίζεται μόνο στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σχέδιο δράσης μας περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων που δεν έχουν σχέση μόνο με τα κρατημέλη μας, αλλά και με δράσεις που πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητες σε διεθνές επίπεδο και αναφέρομαι κυρίως στις ε, συστάσεις που έχουμε κάνει, αποκινούμε το σχέδιο δράσης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί ε, και η φοροαπάτη αλλά και να υπάρξει ενίσχυση ε, των καλών πρακτικών. Αυτό ισχύει βεβαίως και για άλλες χώρες ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών παραδείσων. Αναγνωρίζουμε επίσης ε, ότι προωθώντα αυτές τις αρχές πρέπει να, να προσφέρουμε και μια στήριξη στις χώρες που θα ήθελαν να τηρήσουν αυτά τα πρότυπα αλλά μπορεί να έχουν πρόβλημα ε, δυνατοτήτων για να το πράξουν. Οπότε θα τους δώσουμε τη βοήθειά μας ε, σε αυτές τις χώρες γιατί θέλουμε να τις βοηθήσουμε να μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτές τις αρχές και χρειάζεται μια καλή φορολογική πολιτική για να γίνει αυτό και σωστές, σωστός λειτουργούσες φορολογικές αρχές. Ε, Βεβαίω για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, ή το είπατε κι εσείς, έχουμε μια καλή εμπειρία στον τομέα αυτό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον, στα πλαίσια της οδηγίας για τις αποταμιεύσεις και πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα πρότυπο το οποίο θέλουμε να το διευρύνουμε και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Βλέπουμε κάποια ενθαρρυντικά σημάδια, μηνύματα, ότι αυτό το θέμα συζητάται και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον ΩΣΑ, ως αποτέλεσμα και των συζητήσεων που γίνονται από την ε, πλευρά της Αμερικής σχετικά με τη σχετική πράξη, την ΦΑΤΚΑ, που έχει βέβαια κάποια κενά, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει προωθήσει πολύ το θέμα αυτό της, ανταλλαγής, της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει τώρα διεθνώς μια συζήτηση για τα πρότυπα αυτά και βεβαίως θέλουμε και εμείς να συμβάλλουμε στη συζήτηση αυτή και να προσφέρουμε τη δική μας ευρωπαϊκή εμπειρία στη συζήτηση που γίνεται σε διεθνές επίπεδο. Καλωσορίζουμε λοιπόν την στήριξή σας ε, γι' αυτό και θεωρούμε ότι αυτή είναι μια στήριξη και στην προσπάθεια που θέλουμε να κάνουμε σε διεθνές επίπεδο. Οι, οι συνάδελφοί μου από τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΚ, εγώ είμαι από την ΤΑΞΟΥΤ, υποστηρίζουν ε, τα όσα είπατε για, την, για τις εκθέσεις αναχώρα και τις προσπάθειες για την προώθηση της διαφάνειας σε ό,τι αφορά τα διάφορα ταμεία και τα υπόλοιπα οχήματα. Σταματώ εδώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο Γκάι Σύντομα, Πρόεδρε. Την έχουμε κάνει τη συζήτηση το πρωί ήδη. Αλλά μιλούμε και εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό. Α δούμε τι γίνεται και εκτό Ένωση για το θέμα αυτό. Επικεντρωνόμαστε κυρίω στο μετά, στην εποχή μετά τη. Ε, ε, μετά το, τις, ε, τους στόχους της χιλιετίας. Εγώ στηρίζω την προσέγγιση σας. Ε, πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό και να δούμε πιο πέρα τι θα γίνει. Πρέπει να το δούμε πιο προσεκτικά και πιο σοβαρά. Το είπα και πιο πριν. Κάποιος από το City του Λονδίνου ήρθε να με δει και μου είπε ότι δεν είναι δυνατόν να κάνουμε project accounting για εταιρείες ε, από, που ε, προσπαθούν να εκκαθαρίσουν περιοχές από νάρκες για αποναρκοθέτηση. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας για να μπορέσουμε να προοδεύσουμε στον τομέα αυτό και εγώ γενικώ υποστηρίζω την ε, προσέγγιση σας. Και μια που έχω το λόγο πρόεδρε να πω ότι στο, ε, στο χώρο Γεχούντι Μενοχήν υπάρχει μια, ένας ε, εορτασμός της ε, ημέρας του Αγίου Πατρικίου. Στις 6 και 20. Πριν πάμε στη γιορτή του Αγίου Πατρικίου, να σας πω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για την ομοδότησή μου είναι 21η Μαρτίου στις 18 το απόγευμα. Ψηφοφορία στις 23 Απριλίου. Δεν υπάρχουν θέματα διάφορα. Επόμενη συνεδρίαση, Δευτέρα 22 Απριλίου, από τις 15 με 18 και 30 και Τρίτη 23 Απριλίου από τις 9 μέχρι 12 και 30 και από 15 μέχρι 18 και 30. Αυτά. Σταματούμε εδώ τις, τη συνεδρίαση την απογευματινή της Επιτροπής μας. Σας εύχομαι καλή βραδιά. Καλό βράδυ οι συντονιστές θα συνεχίσουν για μία ωρίτσα. Ναι, είναι αυτό.